Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Ξεκινούμε σήμερα το απόγευμα με το σημείο 14 τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκλήσεις και ευκαιρίες για τα δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα των προσφύγων και τη μεταναστευτική κρίση. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπενιάμ Ντάουιτ Μεσμούρ, πρόεδρο της Επιτροπή των Ηνωμένων για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα απλώ να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση. Νομίζω ότι έχουμε επισκέπτες της κυρίας Φεράρα. Να σας καλωσορίσω θερμά. Πρόκειται για νέου κυρίω ανθρώπου ε, στο πίσω μέρο τη άθουσα. Ε, καλωσορίσατε λοιπόν εκ μέρου και τη κυρία Φεράρα στην επιτροπή μα. Και τώρα να περάσουμε στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μεσμούρ. Εισαγωγικά ε, πριν από την παρουσίασή του, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το Νοέμβριο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία καθόρισε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις συστάσεις στον τομέα αυτό. Έκτοτε έχουν εφαρμοστεί μια σειρά από συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τον περασμένο Μάιο εγκρίθηκε η οδηγία για τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτη ή κατηγορία κατηγορούμενοι σε ποινικέ διαδικασίες από την Επιτροπή μας. Και είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι θα θελήσουν να το συζητήσουν το θέμα αυτό και εδώ σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο και στη συνέχεια αυτού του ψηφίσματος, οι συντονιστές της Επιτροπής Λιμπή αποφάσισαν να καλέσουν τον πρόεδρο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών για να καλύψουμε και τις εσωτερικέ και τις εξωτερικές ψυχέ των πολιτικών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα μέλη επίση τη Επιτροπή, ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προσκληθεί και μπορεί να έρθουν στη διάρκεια τη συζήτηση. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων λοιπόν με τον κύριο Μεσμούρ κατά πάσα πιθανότητα θα μα δώσει μια ευκαιρία να συζητήσουμε τι πιο ε, πρόσφατε εξελίξει ε, ε, ε, στο θέμα αυτό των δικαιωμάτων του παιδιού στα Ηνωμένα Έθνη και το πλαίσιο των ε, προσφύγων και της μεταναστευτικής κρίσης. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Μεσμούρ για την παρουσίασή του και με τα χαράς να ξεκινήσει και η συζήτηση μετά από την παρουσίαση. Παρακαλώ κύριε Μεσμούρ, έχετε το λόγο και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι θα βγούμε κερδισμένοι ε, και οι δύο από αυτή την ανταλλαγή απόψεων και εγώ θα υποφοληθώ αλλά και εσείς θα υποφοληθείτε από αυτά που θα ακούσετε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους παρισταμένους, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διευκόλυναν αυτή τη διαδικασία, κάποιους συναδέλφους από τη UNICEF και άλλες ε, οργανώσεις που ε, βοήθησαν για να γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν θα ήθελα να θεωρήσω τα θέματα δεδομένα, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για την Επιτροπή ε, για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είμαστε 18 8 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και συστήθηκε η Επιτροπή μας βάσει τη σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Όταν ξεκίνησε το 1991 είχαμε μόνο 10 μέλη, αυξήθηκε όμως το έργο της Επιτροπής και επεκτείναμε τον αριθμό των μελών. Τι κάνουμε εμείς ως Επιτροπή. Κύριος ρόλος μας είναι να αναθεωρούμε τις εκθέσεις για τις χώρες και τα 196 κράτη ε, υποβάλλουν εκθέσεις και βάσει των εκθέσεων αυτό ε, αξιολογούμε την κατάσταση των παιδιών και τα δικαιώματά τους στις χώρες αυτές. Οι χώρες ε, υποβάλλουν εκθέσεις όχι μόνο για την πρόοδο που έχουν επιτύχει όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τις προκλήσεις και τι ευκαιρίες υπάρχουν ή θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Η σύμβαση είναι ένα πολύ επιτυχημένο έγγραφο. Πρόκειται για το ε, μόνο έγγραφο που έχει κυρωθεί και από τις 196 χώρες. Και επομένως ε, ε, όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο και του ψηφίσματος που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το Νοέμβριο του 2014 εγκρίθηκε το ψήφισμα και εμείς φυσικά επικροτούμε το περιεχόμενό του. Δεν είναι μόνο η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού βέβαια αυτό που παρακολουθούμε, αλλά παρακολουθούμε και το προαιρετικό πρωτόκολλο για την παιδική πορνογραφία, παιδική πορνεία και την συμμετοχή παιδιού σε ένοπλες σειράξεις. Όπως γνωρίζετε, Υπάρχει και το προαιρετικό ε, πρωτόκολλο, το οποίο ετέθησε ισχύ τον Απρίλιο του 2014 και αυτό το προαιρετικό πρωτόκολλο έχει 29 κυρώσεις και 12 ε, είναι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά τις ε, προσωπικές καταγγελίες. Έχει δημιουργηθεί βέβαια κατάλληλο ε, περιθώριο για τα παιδιά στο μεταξύ σε σχέση με αυτά που είχαμε το 1989 όταν εγκρίθηκε η σύμβαση. Η πρόοδος βέβαια δεν ισχύει για κάθε παιδί. Και τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν ακόμα παιδιά που ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα, παιδιά με αναπηρίες, ε, διακρίσεις, ε, κορίτσια, πρόσβαση στην παιδεία, πρόσβαση στην υγεία. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές προκλήσεις όχι μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και για αναπτυγμένες χώρες. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουμε επισημάνει μετά τον επικοδομητικό διάλογο που έγινε. Ο επικοδομητικός διάλογος συνήθως είναι με μια πολυτεωμαϊκή αντιπροσωπεία η οποία είναι παρούσα στη Γενέβη για να υποβάλει την έκθεση της κάθε χώρας και από εκεί και πέρα ξεκινεί διάλογο με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Συνήθως οι διάλογοι αυτοί ε, διαρκούν για έξι ώρες βάσει της σύμβασης και θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η εφαρμογή της ε, σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού είναι ακόμα εξελίξει. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο, αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη, που εφαρμόζει πλήρω τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών σε όλα τα παιδιά στην επικράτειά τη. Που είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να πω ε, για λίγο. Η έννοια ότι η εφαρμογή τη Σύμβαση δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αλλά όλα τα παιδιά που βρίσκονται εντός της επικράτειας μιας χώρας. Και δεν είναι γιατί το λέω εγώ ή γιατί το λέει η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αλλά γιατί το άρθρο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το προβλέπει αυτό ως υποχρέωση. Πέραν του ρόλου μας ε, για την αναθεώρηση και την εξέταση των εκθέσεων της κάθε χώρας, Έχουμε και προσωπικέ καταγγελίε, οι οποίε ε, λαμβάνονται βάσει του πρωτοκόλλου για τι προσωπικέ καταγγελίε και έχουμε και μια εξέλιξη. Το 2014 έγινε μια συζήτηση για τα δικαιώματα των παιδιών και τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Είναι μια διάσκεψη στην οποία είχαμε διάφορου ενδιαφερομένους και συζητούμε διάφορα τρέχοντα θέματα. Γίνεται κάθε δύο χρόνια και το 2016 έγινε και μια συζήτηση για τα δικαιώματα των παιδιών σε ένα υγιέ περιβάλλον. Και καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν ε, μια σειρά από στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και αφορούν και την κλιματική αλλαγή. Η βασική βέβαια συζήτηση που θα θέλατε να κάνουμε σήμερα αφορά κυρίως το θέμα της μετανάστευσης. Ε, για λόγους οικονομίας χρόνου λοιπόν θα περάσω απευθεία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που θα ήθελα να συζητήσω. Πρώτον, όταν αναφερόμαστε στην μετανάστευση, όπως γίνεται και ε, με όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τη σύμβαση, αναφερόμαστε σε νομικές υποχρεώσεις. Τα κράτη συνειδητά έχουν δεσμευτεί ε, και με τη βούλησή της για αυτά τα σημεία. Και αυτό αποτελεί συγκεκριμένη αφετηρία. Κάθε χώρα, η χώρα από την οποία φεύγουν τα παιδιά, οι χώρες ε, τις οποίες διέρχονται, και στις χώρες στις οποίες αφήκνεται, έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν τα παιδιά. Γι' αυτό σας λέω ότι το άρθρο 2 αναφέρεται σε παιδιά εντός της επικράτειας μια χώρας, όχι που έχουν την ηθαγένεια ή την εθνικότητα μια χώρας. Ξέρω ότι έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις, μας το είπε και ο ε, εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κατά πόσο ε, υπάρχει κρίση ή όχι. Από πλευράς δικαιωμάτων του παιδιού αυτή τη στιγμή υπάρχει κρίση. Υπάρχει κρίση λόγω των αριθμών, υπάρχει κρίση λόγω των παραβιάσεων, υπάρχει κρίση λόγω της ε, βαρύτητας της κάθε παραβίασης και επίσης υπάρχει κρίση διότι οι παραβιάσεις οι οποίες γίνονται συνήθως δεν αφορούν ένα ή δύο δικαιώματα, συνήθως είναι παραβιάσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Και αυτό φυσικά είναι και μία ένδειξη διότι αποτελεί πρόκληση. Ο βασικός λόγος όμως για τον οποίο υπάρχει κρίση και πιστεύουμε ως Επιτροπή ότι πρέπει να γίνει κάτι είναι γιατί δεν είναι αποτελεσματική απάντηση που έχουμε δώσει στη μεταναστευτική κρίση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Και τι εννοώ με αυτό θα σας το εξηγήσω εντός ολίγου. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες διατυπώσεις που δημιούργησαν ε, ε, κάποια προβλήματα για την μεταναστευτική κρίση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μετανάστες που φτάνουν σε μια χώρα χωρίς έγγραφα και μπορεί να βρίσκονται σε ένα νομικό κενό. Εμείς ως ε, Επιτροπή θεωρούμε ότι η αίρια του παράνομος και του μη εγκεκριμένου δεν είναι απαραίτητα επικοδομητική όρη. Ε, και πιστεύουμε ότι παρά το γεγονό ότι αναγνωρίζουμε ότι έχει επιτελεστεί ουσιαστική πρόοδος εντός των κρατών μελών της Ένωσης, η ε, διακριτική μεταναστευτική πολιτική δημιουργεί και την κρίση. Καταρχάς, υπάρχει το εξή θέμα, το θέμα του καθορισμού της ηλικία ενός παιδιού. Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι μια σύμβαση που εφαρμόζεται βάσει ηλικία. Όταν ρωτάμε σε ποιον εφαρμόζεται η σύμβαση, λέμε άτομα κάτω των 18 ετών, εκτό και αν θεωρούνται ενήλικες σε, μικρότερη ηλικία βάσει τη χώρα. Ο καθορισμός της ηλικία, μεταξύ άλλων, ε, γίνεται με συγκεκριμένη ανάλυση. Πρέπει να εξεταστούν τα διάφορα θέματα ε, σε κάθε χώρα. Έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ως Επιτροπή ότι η ε, πρακτική που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή βασίζεται σε μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι και τελικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ίσως και κάποιες μέθοδοι που ε, δεν είναι τόσο παρεμβατικές πριν γίνει ε, ο βιολογικός έλεγχος και η βιολογική ανάλυση. Οι χώρες έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων για κάθε λόγο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουν ξενοφοβία, ρατσισμό, ε, διακρίσεις κλπ. Και θα πρέπει να ξεκινήσουν προγράμματα για να βελτιώσουν την εξοικείωση και να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές απόψεις που υπάρχουν για τους μετανάστες. Όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον, και παρακαλώ σημειώστε τι θα σας πω γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ως Επιτροπή θεωρούμε ότι η σύμβαση των ε, δικαιωμάτων του παιδιού, αν είχε κάποια υποθέματα, θα ήταν ε, τα συμφέροντα του παιδιού να αποτελούν προτεραιότητα. Συχνά συζητούμε με χώρες που έρχονται στην Επιτροπή ε, οι οποίες ε, έχουν πολύ χαμηλές εξελίξεις και ε, ε, εφαρμογή του συμφέροντος του παιδιού. Και μάλιστα αυτό δεν είναι τυχαίο ζήτημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να σκεφτούμε το συμφέρον του παιδιού σε κάθε διαδικαστικό ε, στοιχείο για οτιδήποτε, για την κράτηση των γονιών του, για την επιστροφή, την απέλασή του κλπ. Θα πρέπει στην πολιτική και ε, αυτά τα οποία εφαρμόζονται ε, στην πράξη να λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι το συμφέρον του παιδιού πριτανεύει των υπολείπων. Επομένως, προκειμένου να υπάρχει μια ουσιαστική εφαρμογή αυτού του χαρακτηριστικού του συμφέροντος του παιδιού, η συμμετοχή του παιδιού είναι πάρα πολύ σημαντική. Πώς μπορεί να ε, διαπιστώσει κανείς ποια είναι τα συμφέροντα των παιδιών εάν δεν ακούσουν την άποψή τους. Το δικαίωμα λοιπόν ε, ακρόασης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καθορίσουμε και το συμφέρον του παιδιού. Ε, υπάρχουν ψηφίσματα, οδηγίες, αποφάσεις, πολιτικές, μανιφέστα, ε, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, ε, πραγματικά δεν ξέρουμε αν βοηθούν τα δικαιώματα του παιδιού. Τα υπόλοιπα αφορούν την κατάλληλη τεκμηρίωση, αν υπάρχουν έγγραφα, αν υπάρχουν ταυτότητα, αν υπάρχουν δυνατότητα για επανεγκατάσταση τη οικογένεια, επανένωση τη οικογένεια. Ε, αντιμετωπίζονται ένα σειρά μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δούμε αν υπάρχει εκμετάλλευση, λαθρεμπόριο, τράφικινγκ παιδιών κλπ. Και εδώ έρχομαι στο επόμενο θέμα που είναι η βία κατά των παιδιών και η εμπορία των παιδιών, το τράφικινγκ ασυνόδευτοι ανήλικοι ε, και παιδιά, ε, κυρίως έχουν αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά περιστατικά βίας εναντίον τους. Επομένως, στο βαθμό στον οποίο οι διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Ορισμένες φορές είχαμε σεξουαλική εκμετάλλευση, σεξουαλική κακοποίηση, πολλά παιδιά είναι τραυματισμένα ή με μόνιμες αναπηρίες ε, κατά συνέπεια και επομένως πρέπει να δούμε τι προστασία θα την, τι προστασία θα την χάνουν τα παιδιά και τι καθεστώς θα δίνονται σε αυτά τα παιδιά. Και εδώ έχουμε δύο σχετικά θέματα που αφορούν ε, και την παροχή υπηρεσιών παιδεία και υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Υπήρξε μια έκθεση από τα Ηνωμένα Έθνη, από την ε, Αρμοστία για τους πρόσφυγες, η οποία είχε ως τίτλο Missing Out Refugee Education in ε, Migration Crisis. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία έχει πολλά στοιχεία, δεν θα σας κουράσω με τα στοιχεία αυτά, αλλά ένα από τα βασικά στοιχεία που λέει είναι ότι η βάση της έκθεσης μόνο τα μισά παιδιά μετανάστες πρόσφυγες έχουν πρόσβαση σε παιδεία σε σχέση με το παγκόσμιο ποσοστό που είναι πάνω από 90%. Επομένως η κρίση που αντιμετωπίζουμε για την παιδεία είναι μια κρίση εντός μιας κρίσης. Και ε, επομένως μπορεί να είναι, θεωρηθεί και μια ορολογική, ε, ορολογιακή βόμβα η οποία μπορεί να εκραγεί ανα πάσα στιγμή. Τι ευκαιρίε δίνουμε σε αυτά τα παιδιά, τι συνέχεια θα έχουν αν δεν του προσφερθεί δυνατότητα παιδεία η επανένωση της οικογένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και ξέρω ότι έχουν υπάρξει και κάποια σημαντικά βήματα προόδου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η κάθε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν κάποια κριτήρια ανάλογα με το αν κάποιο είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Αν είναι πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει οδηγία η οποία προβλέπει ε, πολιτης εναρμόνιση στους κανόνες, αλλά η άποψή μας είναι ότι ένας αριθμός από τις οδηγίες ε, προβλέπουν εξαιρέσεις στους γενικούς κανόνες και ενώ κάποιες διατάξεις είναι υποχρεωτικές για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες άλλες είναι προαιρετικές ή δίνουν ε, διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Ως Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εμείς παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά και με επικριτικό βλέμμα τα θέματα αυτά, διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού στα πλαίσια της επανένωσης οικογένεια. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, έρχομαι σε δύο ακόμα σημεία πριν ολοκληρώσω. Το θέμα της κράτηση και της εγγύηση για δίκαιη δίκη εδώ η άποψή μας είναι ότι ε, το καθεστώς μετανάστη ενός παιδιού δεν θα πρέπει να είναι λόγος για την κράτησή του. Η άποψή μας είναι ότι ε, δεν λέμε καν ότι θα πρέπει να είναι ίστατη λύση. Λέμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία μπορεί να προστατεύονται τα συμφέροντα ενός παιδιού βάσει της κράτησής του. Ε, εναλλακτικές λύσεις λοιπόν αντί της κράτησης και να είμαστε βέβαιοι ότι η κράτηση ε, ε, δεν θα πρέπει να γίνεται και θα υπάρχουν δυνατότητες νομιμοποίησης ή απέλασης ενός παιδιού και θα πρέπει να υπάρχει και δικαίωμα ακρόασης σε δικαστικές διαδικασίες για την υποδοχή των γονιών του και επίσης ε, να μπορούν να έχουν και λόγο κατά της κράτησης ή απόλυσης των γονιών τους. Ε, γιατί πρέπει η απόφαση να λαμβάνει υπόψη τους το συμφέρον τους. Και ένα τελευταίο ε, σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το θέμα των εγγυήσεων για μια δίκαιη δίκη και μια έγκαιρη διαδικασία. Εμείς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που ε, αφορά παιδιά θα πρέπει να γίνεται σε ε, ένα τρόπο που θα είναι φιλικό προς τα παιδιά, θα λαμβάνει υπόψη τους το φύλλο των παιδιών και πολλά άλλα στοιχεία και επίσης φρονούμε ότι σε πολλές χώρες προορισμού οι διαδικασίες μετανάστευσης και αποφάσεις δεν ε, γίνονται βάση προδιαγραφών ε, και ε, διαδικασιών που προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Για να υπάρχει λοιπόν δίκαιη δίκη στη διάρκεια των παιδιών, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι, να γνωρίζουν τα δικαιώματα προστασία των παιδιών και επομένω αφορούν και όλου αυτού οι οποίοι δουλεύουν για τα παιδιά και με τα παιδιά. Και φυσικά οι χώρες πρέπει βάσει τη σύμφαση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει κατάλληλη εκπροσώπηση των συμφερόντων του παιδιού, ε, κυδεμόνε με εμπειρογνωμοσύνη σε φροντίδα παιδιών, ε, υπερεθνικέ αρχές που αφορούν προστασία των παιδιών, για να ε, προωθήσουν και τα συμφέροντα των παιδιών. Να ολοκληρώσω, παρά το γεγονός ότι είχα κάποια πράγματα να πω για τα κέντρα υποδοχής και τη φύλαξη των παιδιών. Το βασικό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών. Μπορώ να σας δώσω ένα μακρύ κατάλογο γιατί το λέω αυτό και γιατί έχει αυτή την άποψη η Επιτροπή. Ε, η Επιτροπή προτάθηκε από την Πολωνία και ε, πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν και προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών εντός της χώρας τους αλλά και εκτός της χώρας τους. Και ε, πολλές χώρες εκτός Ευρώπης ε, κοιτούν προς την Ευρώπη για ηγεσία, για καλές πρακτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης κύρωσαν τη σύμβαση χωρίς καμία επιφύλαξη και αυτό ήδη αποτελεί ένδειξη πολιτικής βούλησης. Αλλά το ερώτημα είναι πώς μετρά κάποιος την πολιτική βούληση. Είναι βάση κύρωσης, βάση εκθέσεων, βάση συμμετοχής στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο άλλο εταίρο είναι η Γκρούλακ, ο οποία χρηματοδοτεί την ετήσια διάσκεψη για τα δικαιώματα των παιδιών. Ε, είναι βάση του ρόλου που διαδραματίζουν τα κράτη-μέλη, λοιπόν, ή πολύ πέραν αυτού. Εμείς πιστεύουμε ότι πηγαίνει πολύ πέραν αυτού. Αφορά συντονισμό, σεβασμό των συμφερόντων των παιδιών, ε, καθορισμό των απαραίτητων πόρων ε, και διάθεση αυτών των πόρων και επίσης να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε πολιτική, οποιαδήποτε νομοθεσία έχει στο επίκεντρό της και το θεματολόγιο για τα δικαιώματα των παιδιών. Για παράδειγμα, ε, δεν μπορούμε να συγχωνεύσουμε, για παράδειγμα, το θεματολόγιο για τα θέματα φύλου και τα θέματα των παιδιών. Δεν μπορεί τα δικαιώματα των παιδιών να είναι υποσημείωση. Πρέπει να είναι τμήμα αναπόσπαστο ενός κειμένου τρεις εστάσεις. Πρώτον, πρέπει το συμφέρον του παιδιού να είναι στο επίκεντρο, όχι συλλογικά των παιδιών, αλλά του κάθε παιδιού. Στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής, της νομοθεσίας και της εφαρμογής αυτών των πολιτικών και νόμων. Γνωρίζω ότι έχω αυτή την εξαιρετική ευκαιρία να μιλήσω στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι νομικός και ο νόμος ε, με αφορά ιδιαίτερα, αλλά για τα παιδιά η τήρηση της νομοθεσίας είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι απαραίτητη. Και όχι ε, εξορισμού, αλλά λόγω σχεδιασμού, το άρθρο 4 της Σύμβασης λέει ότι τα κράτη θα λαμβάνουν νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα. Ξεκινά από τα νομοθετικά, γιατί η νομοθεσία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και στην παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Εάν υπάρχει σωστή νομοθεσία, λοιπόν, ε, είναι ε, καταλητικός παράγων για να λαμφθούν υπόψη τα όσα προβλέπει η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν δύο εξαιρετικές ευκαιρίες αυτή τη στιγμή. Η προσεχής έγκριση των ε, νέων αναθεωρημένων καθηγητηρίων γραμμών για τα δικαιώματα των παιδιών στην εξωτερική δράση. Επομένω, εκεί θα πρέπει να στείλετε πολύ στεναρά μηνύματα που αφορούν τα πρότυπα για τα παιδιά, αλλά επίσης και η ευκαιρία να συνεχίσετε από τις βασικές ε, ε, αρχές που υπάρχουν για τα ε, παιδιά και την προστασία τους που παρουσίασε ο Επίτροπος ε, για τα θέματα αυτά το 2016. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά θα πρέπει να γίνουν ευρωπαϊκή πολιτική, ευρωπαϊκό και εκτιμένο. Δύο κανόνες είτε στον τομέα της παιδείας, είτε της υγεία είτε της μεθανάστευσης. Ο πρώτος κανόνας λέει ότι το συμφέρον των παιδιών θα πρέπει να είναι πρωταρχικός παράγον και δεύτερον, πάντα, πάντα, πάντα να θυμάστε τον κανένα παρθυμονέν. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε διάφορους συναδέρφους που θα ήθελα να πάρουν το λόγο. Η κυρία Κινγκακάρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα που ανέφερε και ο κύριος Μέσμουρ. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ να μιλήσετε στην Επιτροπή μας. και που κάνατε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ε, παρουσίαση. Μιλώ και ως ε, μέλος της ε, Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που και ασχολούμαι ιδιαίτερα με τα δικαιώματα του παιδιού στην Υποεπιτροπή αυτή. Αναφερθήκατε στα δικαιώματα των παιδιών κατά τη μετανάστευση. και χαίρομαι που υπογραμμίσατε στο σημείο αυτό την σημασία της εκπαίδευσης για τα παιδιά αυτά, διότι γνωρίζετε ότι περίπου το 50% ε, των 30 ε, ε, χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων είναι παιδιά και των 30 εκατομμυρίων ε, και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην χάσουμε ολόκληρες γενιές επειδή έχουν ε, ε, στερηθεί εκπαίδευσης. Και η μόνη δυνατότητα αργότερα να μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή ή να επιστρέψουν στις χώρες τους και να ξεκινήσουν πάλι μια νέα ζωή. Η μόνη δυνατότητα λοιπόν για να σώσουμε τα παιδιά αυτά από άλλους κινδύνους να τους σώσουμε από τη ριζοσπαστικοποίηση ή του να πέσουν θύματα ε, παιδικής ε, εργασίας ε, ή να χρησιμοποιηθούν σε ένοπλε δυνάμει. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα. Ε, γι' αυτό τα θέματα αυτά συνδέονται μεταξύ του Και το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι αυτό της παιδική εργασία. Έχω ε, κάποια στοιχεία από τον ILO και την Παγκόσμια Τράπεζα. 120 εκατομμύρια παιδιών κάτω της ηλικίας όταν 14 ετών ε, εργάζονται και πολλά από αυτά στις ε, χειρότερες μορφές ε, παιδικής εργασίας με πρακτικές ε, σκλαβιάς ουσιαστικά, με εξανακασμό, σεξουαλική κακοποίηση κλπ. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Πρόκειται και για ένα θέμα που συνδέεται με αυτό που είπατε στην αρχή, την, τα παιδιά στις ένοπλες ε, σειράξεις. 10.000 ε, παιδιά κάτω της ηλικίας των 15 ε, υπηρετούν σε στρατεύματα, σε ένοπλες ομάδες. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Τα θέματα αυτά δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, μας ανησυχούν όμως ε, και ε, αναφέρθηκαν σήμερα στην Επιτροπή μας. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το συμφέρον των παιδιών στο πλαίσιο του διαδικτύου και πώς ε, μπορούμε να τα προστατεύσουμε από τη ριζοσπαστικοποίηση, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους σε, σε περιπτώσεις κυβερνοεκφοβισμού. Εσείς λοιπόν, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τι κάνετε, τι μπορείτε να κάνετε για να πετύχετε πλήρη εφαρμογή της σύμβασης και τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που ε, ε, αποτυχάνει η εφαρμογή της σύμβασης. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις της εργασίας σας. Ευχαριστώ η Ναταλή Κρίσπεκ. Πρωτού να πάρει το λόγο θα ήθελα όμως να την ευχαριστήσω και την ομάδα την ε, Άλτε που κάλεσαν ε, τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, του ΟΗΕ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και ιδιαίτερος να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ για την παρουσία του εδώ στη συζήτησή μας. Και το λέω αυτό γιατί όπως φάνηκε και από την τοποθέτηση τη συναδέλφου Κίν Καγκάλ, τα προβλήματα για τα δικαιώματα του παιδιού είναι πολύ άριθμα, είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και αφορούν όχι μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν χρειάζεται μια συντονισμένη δράση, δυναμική, γιατί οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι, είναι μια υποχρέωση ε, που την έχουμε όλοι από τη φύση και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε το συμφέρον του παιδιού, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι στο κέντρο των αποφάσεων μας είτε πρόκειται για την νομοθεσία είτε οτιδήποτε άλλο. <clears throat> Αναφερθήκατε στο ζήτημα της μετανάστευσης την αύξηση του αριθμού των μεταναστών που εισέρχονται σήμερα στο ευρωπαϊκό έδαφος και αναφέρατε δύο προτεραιότητες κατά την άποψή σας, τις προτεραιότητες που θα έπρεπε να έχει η Ευρώπη ανάμεσα στα εκατοντάδες ερωτήματα που τίθενται βέβαια και θέματα που τίθενται, αλλά ε, αναφέρατε δύο κύριες προτεραιότητες για να δημιουργηθεί μια σωστή πολιτική απάντηση στο θέμα. Θα ήθελα να σας ε, ζητήσω λοιπόν να ε, μου τις εξηγήσετε πιο αναλυτικά. Τώρα θα έρθω σε ένα θέμα που αφορά περισσότερο την ε, Γαλλία, την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Περιού του Φεβρουαρίου του 2016, που ε, διατύπωσε ε, επικρίσεις για μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα την πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη, τη σωματική τιμωρία ή τα παιδιά μετανάστες. Και το ερώτημά μου είναι πώς θα δοθεί συνέχεια και πώς θα συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος με την γαλλική κυβέρνηση μετά από την έκθεση αυτή. Επίσης, όσον αφορά την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας. Θα ήθελα να μου δώσετε και για αυτό το θέμα την άποψή σας ε, και τις προτάσεις σας ως πρόεδρος της Επιτροπής του τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ευχαριστώ κυρία Καταρίνα Τσινίτσι Είναι η επόμενη ομιλήτρια. Να σας ενημερώσω ότι ήταν και η συγγήτριά μας για το θέμα των διαδικαστικών ε, εγγυήσεων ε, στις ποινικέ διαδικασίες για τα παιδιά, που αφορούν παιδιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να καλωσορίσω τον κύριο Μασμούρ, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσίαση και την εισαγωγή που μας έκανε. Να πω ότι ακούγοντάς τον πραγματικά, θα έλεγα για μένα και όχι μόνον, ε, τα λόγια σας ήταν η μουσική στα αυτιά μου. Ε, πραγματικά πιστεύω ως πρόεδρος της ε, κοινοβουλευτικής της ομάδας αλλά και των ε, μελών που συμμετέχουν ε, σεβόμαστε απόλυτα την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων παιδιών. Εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί ε, πολλά χρόνια με το θέμα αυτό πριν γίνω ευρωβουλευτή, και πραγματικά είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι πρέπει η προστασία των παιδιών και το συμφέρον των παιδιών πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών, πέραν βεβαίω και των πολιτικών τη κάθε χώρα. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησα, παρεμβαίνοντα και στην Ολομέλη άλλωστε, στον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς και στην Επίτροπο Γιούροβα, με την οποία συναντηθήκαμε και σε άλλες περιπτώσεις, να θέσουν στο επίκεντρο του θεματολογίου για τη μετανάστευση και την προστασία των ανηλίκων και το ε, συμφέρον ε, των παιδιών. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλά πράγματα και ε, πολλές παρατηρήσεις θα μπορούσα να κάνω, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μωράες ότι υπενθύμησε ότι εγώ είχα την τιμή να ασχοληθώ με την οδηγία για τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τους ανήλικους στις ποινικέ διαδικασίες και συμπεριέλαβα και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου για αυτή την οδηγία που είναι η πρώτη μεταξύ άλλων ε, του τομέα αυτού ε, και συμπεριέλαβα όλες εκείνες τις ε, ε, προϋποθέσεις και τις εγγύησεις στις οποίες αναφερθήκατε, διότι είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι η ποινική διαδικασία πρέπει να βασίζεται στο κάθε παιδί. Όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, η κάθε με περίβασή μας θα πρέπει να αφορά το κάθε παιδί, γιατί κάθε παιδί έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, συγκεκριμένες ανάγκες ε, για κάθε προφίλ, επομένως όταν εμείς νομοθετούμε για τους ανηλίκους πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτή την ιδιαιτερότητα. Για να αναφερθώ και λίγο στην πυλική διαδικασία, ε, Καταρχάς πρέπει να συμμετέχει στην ακρόαση και το παιδί, πρέπει να υπάρχει στήριξη και από ειδικού και από την οικογένειά του, υποχρεωτική νομική αρρωγή κατά τη διάρκεια όλες τις διαδικασίες, ε, ε, οι κυρώσεις ε, θα πρέπει να είναι κυρώσεις ε, για να εκπαιδεύσουν και η ποινή φυλάκισης θα πρέπει να είναι μόνο η εξαίρεση και επομένω και πάντα σε ξεχωριστό σοφρονιστικό κατάστημα το οποίο θα έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικέ ανάγκες των παιδιών. Επομένω πρέπει να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή προσοχή στα παιδιά. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σταθώ και στους ε, ανήλικους μετανάστες που είναι αυτοί που την χάνουν όλη τη προσοχή μα ε, σήμερα και δικαίω. Όσον αφορά του ανήλικου μετανάστε, λοιπόν, εγώ πιστεύω και το είπαμε, οι πολιτικοί και οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη κάθε χώρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη του ότι ο ανήλικο μετανάστε είναι κυρίω παιδί. Ε, μετά είναι παιδί μετανάστευση, αλλά πρωτίστως είναι παιδί. Επομένως, πρέπει να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα προστασίας που αφορούν παιδιά. Για τα ασυνόδευτα ανήλικα θα πρέπει να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη, ε, ε, θεραπείες αν χρειάζονται για θέματα υγείας, να υπάρχει ε, παιδεία, ένταξη. Αυτό από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που φτάνουν στα hot spots. Και από εκεί και πέρα να το συνοδεύουμε πάντα με τη βοήθεια ειδικών βεβαίω και την υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων που στον τομέα αυτό, όπως και σε άλλους, αλλά στο συγκεκριμένο τομέα δίνουν εξαιρετική συνεισφορά στα θεσμικά όργανα, να τα συνοδεύουμε στην όλη τους πορεία. Και ολοκληρώνω για να δώσουμε και περιθώριο να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Για τους ασυνόδευτους ανηλίκους υπάρχει η εξής δυσκολία η οποία πορεύει από το γεγονός ότι πολλοί ε, από αυτούς είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Είναι οι λεγόμενοι ανήλικοι οι οποίοι εξαφανίζονται. 10.000 ήταν πέρσι, άλλοι τόσοι φέτος και ήδη στη χώρα μου στην Ιταλία που πιστεύω ότι έχει εφαρμόσει νομοθεσία για την προστασία των παιδιών σε πολύ αυξημένο επίπεδο, έχουμε ήδη 5.000. Επομένως είναι πολύ αυξημένος ο αριθμός. Και αυτό συχνά προκύπτει από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητά τους σωστά δεν ξέρουμε ποιοι είναι και επομένως αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Διότι αν δεν μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητα ενός παιδιού, σίγουρα δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε από εκεί και πέρα στις μετακινήσεις του. Και θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας επ' αυτού και ολοκληρώνω ευχαριστώντας σας για την παρουσία σας εδώ. Πιστεύω ότι αυτό είναι θεμελιώδου σημασία. Να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε σωστά την ταυτότητα ενό παιδιού για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τι μετακινήσει του στη συνέχεια και μετά να το προστατεύσουμε και να αποφύγουμε να αντιμετωπίσει κινδύνου εκμετάλλευση να καταλήξει στο οργανωμένο έγκλημα όλους αυτούς τους πολύ αυξημένους κινδύνους που δυστυχώς ε, αντιμετωπίζουν ιδίως τα πιο μικρά παιδιά. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω και την άποψή σας γι' αυτό. Και κάτι τελευταίο. Η 25η επέτειος της σύμβασης ε, του ΟΗΕ οδήγησε εμένα και σε κάποιους άλλους συναδέλφους να ζητήσουμε ένα ψήφισμα στο οποίο ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσει τη σύμβαση, να την κυρώσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να ε, εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να γνωρίζω την άποψή σας επ' αυτού. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Alahago, please. Thank you, Chairman. I have two questions to Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει έχω προς τον κύριο Μεσμούρ. Στη χώρα μου, τη Φιλανδία, πάνω από το 70% των ετούντων άσυλο που ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι αποδεικνύεται ότι είναι άνω των 18 όταν εξεταστούν. Ε, δύο χρόνια έχουμε περιθώριο λάθους, ε, οπότε ο πραγματικός ε, αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος και αυτοί είναι απλά οι άνθρωποι που ε, υφίστανται τέτοιες εξετάσεις, αυτοί δηλαδή που ισχυρίζονται, ε, αυτοί που φαίνεται να ε, είναι μεγαλύτεροι από την ηλικία που ισχυρίζονται ότι έχουν. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία κατάχρηση του, της έννοιας του ασυνόδευτου ανηλίκου που προκαλεί υποψία και κινησμό στο κοινό και γι' αυτό ε, η εξέταση για τον καθορισμό της ηλικίας ε, αποτελεί σημαντικό εργαλείο ώστε να προστατεύσουμε ε, αυτούς που πραγματικά είναι παιδιά και που πράγματι χρειάζονται προστασία. Από τις αρχικές σας παρατηρήσεις δεν κατάλαβα τι, ποια είναι η δική σας θέση όσον αφορά τις εξετάσεις για τον καθορισμό της ηλικίας. Τι προτείνετε εσείς. Και άλλη μία ερώτηση. Φαίνεται να είστε κατά της κράτησης ανηλίκων υπό οποιασδήποτε περιστάσεις. Υπάρχουν όμως εκατοντάδες ανήλικοι ε, ετούντες άσυλο που έχουν εξαφανιστεί. Ο Θεός ξέρει πού, πού βρίσκονται. Αυτοί των οποίων οι αιτήσει ε, απορρίπτονται, εξαφανίζονται ε, ασχέτως ηλικίας. Αυτό δεν είναι προς ε, συμφέρον ε, κανενός ούτε του ιδίου του ενδιαφερόμενου. Πώς ε, προτείνεται να αποτρέψουμε τέτοιες εξαφανίσεις χωρίς κράτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει μετάφραση από τα φιλανδικά σήμερα. Έπρεπε να έχω κάνει τη σχετική διευκρίνηση στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης. Εν πάση το αναφέρω επισήμως τώρα. Ζήτω συγγνώμη. Η Κορνίλια Έρνστ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλόντ. Ε, είπατε ότι σε καμία χώρα του κόσμου δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως ε, η σύμβαση του ΙΕ. Αναφέρατε πολλά παραδείγματα και είπατε ότι πρέπει να αποτελέσει οριζόντιο καθήκον ε, η υπεράσπιση των ε, δικαιωμάτων των παιδιών. Αλλά τα δικαιώματα των παιδιών δεν μπορούμε να τα ε, διαχωρίσουμε από τα γενικά δικαιώματα. Τα παιδιά ανήκουν σε μια οικογένεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς βλέπουμε τα δικαιώματα της οικογένειας. Ε, συμφωνώ τους μαζί σας ότι δεν επιτρέπεται να κρατούνται τα παιδιά. Βρίσκω εξωφρενικό να το σκέφτεται κανείς ε, αυτό, να βάλει τα παιδιά στη φυλακή. Φυσικά, συμφωνούμε με τη θέση αυτή ότι τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν φυλακή. Αλλά ούτε και οι γονείς έτσι δεν είναι. διότι αυτά τα δύο θέματα συνδέονται μεταξύ τους ε, και γενικά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς αντιμετωπίζουμε τους ετούντες άσυλο, τους πρόσφυγες. Το παιδί σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και το γενικότερο πλαίσιο. Αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ, διότι νομίζω ότι ούτε και οι ενήλικες πρέπει να πηγαίνουν φυλακή, εκτός βέβαια να έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα, οπότε είναι τελείω διαφορετική περίπτωση. Ένας ε, συνάδελφος είπε ότι έχουν εξαφανιστεί πολλά παιδιά. Ε, εξαφανίστηκαν στην έρημο, μερικά ε, έχουν ε, χρησιμοποιηθεί για εμπόριο οργάνων ε, στο κοσυφοπαίδιο. Η ερώτησή μου είναι τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ε, τον τρόπο να υπάρχει νόμος τρόπος σόδου στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επόμενο θέμα που με ενδιαφέρει εμένα είναι η οικογενειακή επανένωση. Ξέρουμε ότι πολλά παιδιά από το Αφγανιστάν ή από αφρικανικές χώρες ταξιδεύουν ασυνόδευτα και τίθεται το θέμα αργότερα της οικογενειακής επανένωσης. Στη Γερμανία και σε άλλες ε, χώρες γίνονται προσπάθειες μετά για επανένωση. Μπορείτε να πείτε λίγα λόγια για το θέμα αυτό. Τι θα ήταν σημαντικό να ρυθμίσουμε στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα αυτό. Τρίτον, είπατε Ε, χρειαζόμαστε ειδικό προσωπικό για τα παιδιά μεταναστών. Τι ακριβώς εννοείτε στα hot spots, ε, στα διάφορα ιδρύματα να έχουμε επιπλέον προσωπικό, επιπλέον ρυθμίσεις, κανόνες ε, για τα παιδιά, για την προστασία των παιδιών δηλαδή ή έχετε άλλες προτάσεις. Θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Χαίρομαι για την παρουσία σα εδώ και τη δυνατότητα που έχουμε να συζητήσουμε το ζήτημα των δικαιωμάτων του παιδιού. Έχω πολλά ερωτήματα και τα κυριότερα είναι συγκεκριμένα. Τώρα βεβαίω μπορεί να μην έχετε όλες τις απαντήσει. Ε. Αλλά θα τα θέσω. Έχετε στα χέρια αριθμητικά στοιχεία για τον αριθμό των παιδιών που ήταν ε, ε, ξεριζώθηκαν από τις αιστείες τους και έχουν πέσει θύματα της εμπορίας ανθρώπων και των εγκληματικών δικτύων. Γιατί το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και ακόμα περισσότερο των παιδιών μεταναστών είναι ένα θέμα στο οποίο μας έχει απασχολήσει πρόσφατα και στο οποίο έχουμε ε, υποβάλει προτάσεις. Δεύτερο θέμα, προσπαθώντας να κάνουμε τον απολογισμό τον, κάτι, ε, της κατάστασης των δικαιωμένων των παιδιών. Υπάρχουν χώρες, υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες να συνεχίζουν να ε, επιλέγουν την οδό της κράτησης ανηλίκων υπάρχει αύξηση ή μείωση αυτών των χωρών και μήπως έχουν προταθεί ε, εναλλακτικέ λύσεις. Τρίτο ερώτημα. Ε, η κατάσταση στη Συρία ε, και η έρευνα που έγινε για τα παιδιά που βρέθηκαν στην Τουρκία και εξαφανίστηκαν. Εάν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτό, και αν υπάρχουν πρωτοβουλίε σε παγκόσμιο επίπεδο που θα μπορούσαν να αναλυφθούν έτσι ώστε ε, να σταματήσει η εκμετάλλευση των παιδιών από εμπόλεμε περιοχέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βίνπερκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σα ευχαριστώ για τι πληροφορίε που λάβαμε εδώ σήμερα. Το άρθρο 54 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού λέει ότι όλα τα παιδιά μέχρι ε, την ηλικία των 18 ετών έχουν ε, τα ίδια δικαιώματα. Ε, το συμφέρον του παιδιού ε, και τα δικαιώματα του παιδιού είναι δύο γενικές αρχές που διέκουν το σύνολο της σύμβασης ε, και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανη που η Σουηδία προσπαθεί να εφαρμόσει πλήρως την σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Θα αναφερθώ στην μεταναστευτική κρίση που επηρέασε πάρα πολύ την Σουηδία, ιδιαίτερα όσον αφορά συνόδευτους ανήλικους. Η Σουηδία έχει πληθυσμό σχεδόν 10 εκατομμύρια ε, ανθρώπους ε, και υποδεχτήκαμε 35.000 ε, ασυνόδευτους ανηλίκους. Αμφισβητείται στην Σουηδία η ηλικία των παιδιών αυτών και μάλιστα παιδίατρος στη Σουηδία είπε ότι Κάποια από αυτά τα δίθεν παιδιά είναι μέχρι ε, και 40 ετών και δεν ε, κάνουμε εξετάσεις για το καθορισμό της ηλικίας. Ε, καταχωρίζουμε την ηλικία που ισχυρίζονται οι ίδιοι ότι έχουν, το οποίο σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Πολλά από αυτά τα αγόρια ή αυτοί οι νέοι άνδρες Ε, υποτίθεται ότι έχουν ηλικία 15 έως 17 ετών ε, και επίσης 11 ε, τέτοιοι είναι οι άντρες, αντιστοιχούν σε κάθε κορίτσι. το θέμα λοιπόν είναι ότι μιλάμε για το συμφέρον των παιδιών. Θα πρέπει λοιπόν ενήλικοι άντρες να κλέβουν ε, πόρους που προορίζονται ε, για παιδιά. Νομίζω ότι έτσι παραβιάζουμε την ε, σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών. Ρωτώ λοιπόν, δεν πιστεύετε και εσείς ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η εξέταση για τον καθορισμό της ηλικίας, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ακριβώς τα παιδιά και οι πόροι που έχουμε προβλέψει για τα παιδιά να ε, πηγαίνουν πράγματι στα παιδιά και όχι σε νέους άντρες. Ευχαριστώ. κυρία Φεράρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον κύριο Μέσλουν. Εγώ είμαι εισηγήτρια για την πρόταση κανονισμού για τις ε, κοινέ διαδικασίες ασύλου. Και στα πλαίσια της πρότασης Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία αφορούν ε, τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Υπάρχει υποχρεωτική νομική προστασία, ε, ένας κηδεμόνας το συντομότερο δυνατόν ε, μετά από πέντε εργάσιμες ημέρες το αργότερο από την άφηξη του παιδιού και επίσης για κάθε κηδεμόνα δεν μπορεί να υπάρχει δυσανάλογος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων, κάτι το οποίο είναι θετικό ε, να σας δώσω το παράδειγμα της Ιταλίας. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες ε, για κάθε κυδεμόνα ε, έχουμε περίπου 70 συνόδευτους ανηλίκους. Επομένως πρόκειται για μια σχέση την οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί. Υπάρχει επίσης και κατάλληλο σύστημα ελέγχου για τις παροχές αυτού του κηδεμόνα εντό εισαγωγικών. Και όλα αυτά τα οποία σας είπα είναι θετικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας του 2013 και επομένω ε, και του μελλοντικού κανονισμού. Υπάρχουν όμως και κάποιες πτυχές ε, οι οποίες ε, μας δημιουργούν αμφιβολίες και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμοί στις ε, ε, ταχείες διαδικασίες, διαδικασίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και σε περιορισμό της ε, προσωπικής ελευθερίας. Το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε ε, χρήση αυτών των ε, διαδικασιών και όχι εξαίρεση για τα συνόδευτα ανήλικα παιδιά ε, μας δημιουργεί αμφιβολίες. Για παράδειγμα, αυτή η ταχεία διαδικασία εφαρμόζεται όταν αποφασίσουμε ότι ένα ανήλικος ε, φτάνει από μια ασφαλή ε, χώρα και από εκεί ξεκινά η ταχεία διαδικασία. Θα ήθελα όμως να ακούσω και την άποψη τη δική σα ε, για το θέμα αυτό, για τη συγκεκριμένη αυτή πτυχή, όπω επίση και για την ιατρική εξέταση προκειμένου να καθορίσουμε την ηλικία του ανηλίκου. στην πρόταση του κανονισμού προβλέπονται κάποιες συγκεκριμένες εγγυήσεις και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι δεν μπορεί να υποχρεωθεί ένας ανήλικος να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση για τον καθορισμό της ηλικία του. Ταυτόχρονα όμως η άρνηση από πλευράς ανηλίκου μπορεί να ε, θεωρείται ότι ε, είναι υπόθεση ε, ότι είναι ενήλικος. Ε, Ξεκινούμε δηλαδή από μια υπόθεση ότι είναι ενήλικας ο ανήλικος όταν αρνηθεί την ιατρική εξέταση. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας και από αυτού, κυρίως όσον αφορά το συμφέρον του παιδιού. Και επίσης ε, δύο ακόμα πτυχές οι οποίες ε, απορρέουν από την πρόταση κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου. Η πρώτη αφορά κάτι το οποίο ζήτησε ήδη ο συνάδελφος ε, Αλάχο επειδή υπάρχει όλο ένα και αυξανόμενο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που εξαφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, τι προτείνετε εσεί προκειμένου να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίζουμε τέτοιε εξαφανίσει. Ε, για πρακτικού λόγου, ε, τι θα μπορούσαν να κάνουν τα κράτη-μέλη από πρακτική σκοπιά, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει το κάθε κράτο μέλο. Και επίση, όσον αφορά την πτυχή τη υποδοχή. Και εδώ θα σα δώσω το παράδειγμα τη Ιταλία. Έχουμε διάφορα σκάφη τα οποία φτάνουν και υπάρχουν διάφορες ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι δήμαρχοι των δήμων που υποδέχονται αυτούς τους ε, αλλοδαπούς ασυνόδευτους ανηλίκους αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες από πλευράς ε, και επιμελητίας αλλά και από πλευράς οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων. Δεν υπάρχουν ε, χώροι κατάλληλοι για την υποδοχή αυτών των ανηλίκων και πολλές φορές καταλήγουν να στεγάζονται σε αθλητικά κέντρα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλος χώρος να στεγαστούν και ε, είναι όμως η μόνη λύση επειδή δεν υπάρχουν άλλες. Ε, όπως επίσης ε, και όσον αφορά την παιδεία αυτών των παιδιών. Όταν αναφερόμαστε σε ανηλίκους, αναφερόμαστε σε ε, παιδιά κάτω των 18 ετών και κάτω των 16 βεβαίως και μεταξύ αυτών υπάρχουν και παιδιά τα οποία χρειάζονται να κάνουν μαθήματα για να μάθουν γράμματα γραφή και ανάγνωση και το να υπάρχουν ε, κρατικοί πόρου ε, για την ε, διδασκαλία παιδιών των, κάτω των 16 ετών αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί το να βάλουμε ένα 16χρονο ή 17χρονο παιδί μαζί με παιδιά δημοτικού στο σχολείο δεν θεωρείται λογικό. Επομένως υπάρχει πρόβλημα και με ανελίκους οι οποίοι είναι μεταξύ 16 και 18 ετών γιατί δεν μπορούμε να τους εγγυηθούμε ότι θα μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοια μαθήματα γραφής και ανάγνωσης είναι λοιπόν πρακτικό το ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε κατάλληλη υποδοχή αυτών των παιδιών και να σεβαστούμε και τη σύμβαση ε, για τα δικαιώματα του παιδιού. Ευχαριστώ. Thank you. And finally, Thomas please. Ευχαριστώ και κλείνουμε τον κύριο Δεν θα με γιατί βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσει. Κάποια πολύ σύντομα ερωτήματα θα πέσω. Σας ευχαριστώ κύριε Μεσπούρ για την παρουσία σας εδώ. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού συχνά αποτελεί αντικείμενο κριτικής, ε, επικρίνεται από χώρες ε, όχι μόνο της ε, Ευρώπης. Έχω ακούσει επικριτικά σχόλια από το Λίβανο, από χώρες της Αφρικής και ο λόγος που σας ασκείται αυτή η κριτική είναι επειδή η Επιτροπή του ΟΗΕ ε, είναι ιδιαίτερο αυστηρή με τις φτωχέ χώρες και δεν επιδεικνύει την ίδια ευστηρότητα με πλουσιότερες αναπτυγμένες χώρες. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Νορβηγία. Εκεί έγιναν διαδηλώσεις. Ε, υπάρχει μια νέο μαρξιστική οργάνωση ναι, η οποία έχει συστηματικά καταστρέψει οικογένειες. Και δεν έχετε επικρίνει αυτή την πρακτική. Τα παιδιά μεταναστών, κυρίως Αφρικανών μεταναστών, ε, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους, τα, τα, τα αποκόπτουν από την οικογένειά τους ε, με αυτές τις διαδικασίες. Και ε, αυτό επειδή, για παράδειγμα, οι γονείς τους δεν δουλεύουν. Θα ήθελα να μου ε, εξηγήσετε ποια είναι η θέση της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Ε, επίσης, για το ζήτημα της Γαλλίας, για την ε, κατάσταση στο Καλέ ή την ε, γεγονό ότι επέτρεψε η Γαλλία να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές και να βρεθούμε με έναν καταβλισμό στον οποίο εκατοντάδες παιδιά έχουν υποφέρει και έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Επιπλέον, έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, για παράδειγμα στην ε, Σερβία. Και έχω ακούσει μαρτυρίες ανθρώπων που μου κατήγγυλαν ότι ερχόντουσαν ε, πλούσιοι μετανάστες, οι οποίοι έρχονταν και αγόραζαν παιδιά, ε, παιδιά μεταναστών, με τιμές που κυμαίνονταν κοντά στις 5.000 ευρώ, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μεγαλύτερε πιθανότητες να του δοθεί άσυλο στην Ευρώπη. Και δεν έχω διαβάσει πουθενά η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού το έχει επικρίνει αυτές τις ε, καταστάσεις. Πολύ θα ήθελα να με διαψεύσετε. Ο πρόεδρο, πράγματι δεν περίμενα τόσες πολλές ε, και ενδιαφέρουσες ε, και λεπτομεριακέ ερωτήσει να θέσουν οι συνάδελφοι. Αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον τους για τα θέματα αυτά είδα ότι κρατούσατε ε, σημειώσεις, είδατε επίσης ότι το ζήτημα της Συρίας αναφέρθηκε πολλές φορές από τους συναδέλφους που δείχνουν το ενδιαφέρον τους. Έχετε το λόγο για να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλες τις ερωτήσεις. Με βλέπετε, χαμογελώ. Διότι δείχνει το ενδιαφέρον σας δείχνει ότι αντιμετωπίζετε πρακτικά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης, αλλά ότι θέλετε να τα αντιμετωπίσετε όσο γίνεται πιο σύντομα. Έχω σημειώσει λοιπόν τις ε, ερωτήσεις. Ο πρόεδρος μου είπε ότι έχω περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή μου. Ε, όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, ότι επιλέγουμε ως Επιτροπή με ποιους συνομιλούμε. Ε, υποθέτω ότι θέλετε ε, να πω ότι έχετε άδικο. Διαφωνώ με την εκτίμησή σας. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαμε ιδιαίτερα επικριτική δήλωση όσον αφορά τα παιδιά στο καλέ. η πολιτική και όσον αφορά την πολιτική διαμάχη ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Έχουμε επίσης ε, δημοσίευσει δηλώσεις για την Αυστρία, ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 1,5 χρόνο για την ε, μεταναστευτική κρίση, για παράδειγμα. Για να σας δώσω μια εσωτερική ματιά, ως Επιτροπή κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα ε, στο πότε πρέπει να φωνάζουμε, πότε πρέπει να ψιθυρίζουμε. Μερικές φορές ε, στέλνουμε επιστολές ε, χωρίς να τις δημοσιεύουμε. Κάποιες χώρες που εκπροσωπούνται εδώ έχουν λάβει επιστολές. Για παράδειγμα, σχετικά με νομοσχέδια στο Κοινοβούλιο για την, χρήση, την εκμετάλλευση των παιδιών στην επαιτία και είπαμε ότι μπορεί, για παράδειγμα, να, είναι, ε, να δημιουργούν διακρίσεις επειδή στοχεύουν ειδικά στα παιδιά των Ρωμά. Ε, δεν ε, θα αναφερθώ πάλι σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά στείλαμε και πάλι επιστολή σχετικά με την μεταχείριση παιδιών με αναπηρίες σε κάποια χώρα. Με άλλα λόγια, όλες τις χώρες, από το Αφγανιστάν στη Ζιμπάπουε, από το Α μέχρι το Ζ, ε, τις ε, αντιμετωπίζουμε ίσα. Και αποφασίζουμε ε, αν θα φωνάξουμε ή αν θα ψιθυρίσουμε ή αν απλά θα συνομιλήσουμε μαζί τους. και ε, ακούστηκαν πράγματα για την παιδική εργασία, για ε, τα παιδιά στις ένοπλες σειράξεις. Ε, συμφωνώ απολύτως. Το βασικό ερώτημα όμως ήταν τι γίνεται με την εφαρμογή, την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών και ιδιαίτερα τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Το βασικό θέμα εδώ είναι η πολιτική βούληση και πώς την μετράμε με την κύρωση των συμβάσεων ε, ή με γενικότερα θέματα, ε, το τι μπορεί διατίθενται, να φροντίσουμε οι οργανώσει της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία ε, χωρίς να βασιζόμαστε υπερβολικά στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για κάποιες βασικές υπηρεσίες. Η σύμβαση απαιτεί νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα και πολλά κράτη-μέλη βασίζονται πάρα πολύ στα νομοθετικά μέτρα. Έρχονται λοιπόν και μας λένε ότι έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία για την, ε, για την εμπορία ανθρώπων, ε, για την παχυσαρκία, για διάφορα θέματα. Ε, αλλά εμείς δεν θέλουμε να πούμε ότι τα λέτε ωραία, θέλουμε να πούμε ότι τα κάνετε καλά. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι πόρους έχετε διαθέσει, το ανθρώπινο δυναμικό σας, ε, κατά πόσο το έχετε ενισχύσει η νομοθεσία, ε, η πολιτική και η πρακτική αξιολογούνται εκ των υστέρων. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές προκλήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες. Ο συντονισμός αποτελεί σημαντική πρόκληση, όχι μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και για τις αναπτυγμένες. Σε διάφορες περιπτώσεις ε, χρειάστηκε να καταστήσουμε σαφές ότι ε, τα δικαιώματα των παιδιών είναι θέμα οριζόντιο και ότι θα πρέπει ε, οι αλλαγές να γίνουν κοντά σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Έχουμε δει αποδυναμωμένο συντονισμό, κατακαιρματισμό. Και σε διάφορες περιπτώσεις τα παιδιά χάνονται στα νομοθετικά κενά. και παρεμβαίνουμε μόνο εάν διαπιστώσουμε ότι κάποια ρύθμιση οδηγεί σε παραβίαση των, ανθρώπων, ε, των, των δικαιωμάτων των παιδιών. Ε, δεν, θα αναφερθώ πάλι, δεν, θα, δεν θα αναφέρω πάλι το όνομα συγκεκριμένου κράτους μέλους, ε, αλλά ε, επειδή η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν θέμα ε, των περιφερειών, ενώ η δευτεροβάθμια ήταν θέμα ε, ε, της Ομοσπονδιακής ε, Κυβέρνησης, πολλά παιδιά δεν προχωρούσαν από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό τονίζω πάλι ότι θα πρέπει ότι παραμένει σημαντικό θέμα το πώς μπορούμε τα δικαιώματα των παιδιών να αποτελούν το σημείο εστίασης κατά την νομοθεσία και κατά την λήψη μέτρων. Ε, τα παιδιά είναι, το ότι τα παιδιά είναι μικροί άνθρωποι με μικρά δικαιώματα είναι πεπαλαιωμένη νοοτροπία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Ευρωβουλευτής από τη Γαλλία τρεις προτεραιότητες. Ε, είπε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν ε, στο πλαίσιο της κρίσης της μεταναστευτικής. Ε, σας ευχαριστώ γιατί, πολύ για την ερώτηση αυτή. Με κάνει να χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί, διότι δεν είναι η Ευρώπη η μόνη η Ήπειρος που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω μετανάστευσης. Μάλιστα, εάν κοιτάξετε τους αριθμούς, άλλες περιφέρειες, άλλες Ήπειροι ε, αντιμετωπίζουμε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς και πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από τη Ευρώπη. Δεύτερον, η μεταναστευτική κρίση που βλέπουμε εδώ στην Ευρώπη θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να αποτελεί σύμπτωμα. Η κρίση δεν ξεκίνησε το 2014 το 2015. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού δίνει συστάσεις στα κράτη-μέλη ε, από το 1991 Έχουμε μιλήσει για τη μη ένταξη των παιδιών μεταναστών, ε, την, ε, τις διακρίσεις εις βάρος παιδιών που αιτούνται άσυλο. Έχουμε μιλήσει για τα μέτρα για την ασφάλεια που δεν αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Η κρίση λοιπόν δημιουργήθηκε λόγω προηγούμενων κενών ε, στο σύστημα. Ε, κενά όσον αφορά την κυδαιμονία, τα κέντρα υποδοχής ε, κλπ. Έτσι λοιπόν έγινε κρίση επειδή υπήρχαν διάφορα κενά στο σύστημα. Όσον αφορά τις τρεις προτεραιότητες, ως Επιτροπή δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε διάφορα προβλήματα, αλλά ε, υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται και πιστεύουμε ως Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει ε, να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής για να προστατεύσει όλα τα παιδιά που μεταναστεύουν. Θα πρέπει να είναι πλήρες και συγκεκριμένο, να είναι δηλαδή κεντρικό και να έχει την ε, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο κέντρο της. Ε, το άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο ρόλος που παίζετε εσείς στην εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντικός για να αντιμετωπιστεί η παρούσα μεταναστευτική κρίση. Εγώ ε, προέρχομαι από την Αιθιοπία, συνεργάζομαι με την Αφρικανική Ένωση ε, συχνά και αυτή τη στιγμή ε, γίνεται συζήτηση σχετικά με την συνεργασία ε, και για θέματα μετανάστευσης, για παράδειγμα από το, τη Σενεγάλη, το Μαλή, την Νιγηρία, τον Νίγηρα και τη χώρα μου την Αιθιοπία. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ε, σημαντική ευκαιρία αν γίνει σωστά. Δεν ε, έχει κανείς δεύτερη ευκαιρία να κάνει μια καλή πρώτη εντύπωση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ε, κεντρικό ρόλο στη διαδικασία να παίζουν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών και να οικοδομήσουμε στις εμπειρίες που ε, είχαμε ανάμεσα στην ε, Ελλάδα και την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι αυτές τις πρακτικές μπορούμε να τις αντιγράψουμε ε, στην Αφρικανική Ήπειρο. Πάντως νομίζω ότι όλα αυτά θα αποτελούσαν καλό σημείο κίνησης και τελικά θέλουμε ε, να προωθήσουμε την ε, ασφαλή μετανάστευση και νομίζω ότι αυτός ε, είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα πρέπει να δούμε τη μετανάστευση όχι μόνο ως πρόκληση αλλά και ως ευκαιρία. Και πολλοί από εσά θα έχετε ακούσει εδώ ότι εάν το δούμε ως ευκαιρία θα έχουμε και κέρδος. Όσο περισσότερα παιδιά βλέπουν να παραβιάζονται τα δικαιώματά τους, τόσο διαιωνίζεται το πρόβλημα. Τα παιδιά αυτά θα αποτελέσουν πρόβλημα ασφαλείας ε, και άλλα προβλήματα ε, στο μέλλον. Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση για την παιδική πορνογραφία και ε, το διαδίκτυο. Ως Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Παιδιών εξετάζουμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά. Υπάρχουν ε, χώρες που ε, λένε ότι εμείς είμαστε εντάξει, εμάς ο πολιτισμός μας ε, δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε χώρα υπάρχουν προβλήματα παιδικής πορνογραφίας, παιδικής πορνείας και κυβέρνο εκφοβισμού. Είχαμε λοιπόν συζήτηση για τα δικαιώματα του παιδιού στα ψηφιακά μέσα και έχουμε δώσει αναλυτικές κατευθυντήρες γραμμές. Ε, θα πρέπει να έχουμε ε, προγράμματα ευαισθητοποίησης, ε, κατάρτισης και υποστήριξης για, την, για τις ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Όλα αυτά είναι σημαντικά και στο διαδίκτυο και εκτός. Και Γι' αυτό παραμένει και επίκαιρη σύμβαση παρότι υιοθετήθηκε πριν 26 χρόνια. Δεν αναφέρει την λέξη διαδίκτυο, αλλά ούτε το AIDS αναφέρει, ούτε τη ε, την ε, σωματική τιμωρία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εξετάσουμε και το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στο θέμα αυτό, διότι αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα είδαμε σε κάποιες χώρες. Η υλικό πορνογραφίας όταν ε, βρίσκεται στο διαδίκτυο, ο πάροχος ε, των ε, ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος απλά να το κατεβάσει. Βοηθάει αυτό πιθανότατα, αλλά είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει. Όχι, σημαντικό είναι να το αναφέρει κανείς στις αρχές, να γίνει έρευνα. και ε, αυτοί που ε, παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού να ε, λογοδοτήσουν. Θέλουμε να αποφύγουμε την βλάβη στα παιδιά και με τη χρήση των bitcoins. Είδαμε κάποια παραδείγματα. Είχαμε έναν άντρα στι Ηνωμένε Πολιτείε που είχε ένα κορίτσι στο μπάνιο του, έπαιρνε φωτογραφίε και κατάφεραν να κάνουν zoom σε ε, ένα βαζάκι με φάρμακο στην τουαλέτα του και βρήκανε ε, τα πρώτα γράμματα του ονόματός του και έτσι κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Και μάλιστα από την φωτογραφία αυτή ε, μπόρεσαν να βγάλουν και δαχτυλικά αποτυπώματα. Κάτι που απέτησε χρόνο, απέτησε όμως και συνεργασία από πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς. Υπάρχουν λοιπόν πολλά υποσχόμενες εξελίξεις, απαιτούν όμως συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Ο Ιταλός ανέφερε ε, ε, η Ιταλίδα Ευρωβουλευτή ανέφερε την φυλάκιση ως ε, ίστατο μέτρο και τι θα κάνουμε με τους εξαφανιστέντες. Και αυτό είναι θέμα που έθεσαν και άλλοι ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Η δουλειά μα πάνω στη μεταναστευτική κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε αρχές και στα δικαιώματα. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι το διεθνέ δίκαιο δεν είναι δίκαιο. Δεν αποτελεί νομοθεσία. Και λένε γιατί. Λένε διότι δεν υπάρχει μηχανισμός ε, επιβολής. Ε, δεν λένε το ίδιο όμως για το ποινικό δίκαιο, διότι και στο ποινικό δίκαιο υπάρχουν προβλήματα ε, εφαρμογής. Επιβολή του νόμου. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από τις αρχές, από τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει ως κράτη. Και οι δυσκολίες στην εφαρμογή δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε εκπτώσεις στις υποχρεώσεις μας. Αυτό ήθελα να πω. Ε, και όπως είπα νωρίτερα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι τα μόνα που αντιμετωπίζουν μεταναστευτική κρίση. Όσον αφορά την κράτηση ε, ανηλίκων, δεν θα πρέπει ποτέ να κρατούνται για τους σκοπούς ε, ελέγχου της μετανάστευσης. Ε, λέμε ότι δεν δικαιολογείται η κράτηση ε, αποκλειστικά επειδή πρόκειται για συνόδευτό ανήλικο, επειδή έχει καθεστώς μετανάστη ή πρόσφυγα. Έχουμε την ε, στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης 2016-2021, όπου λέει ότι πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια να ε, τερματιστεί η κράτηση παιδιών. Και υπάρχουν παραδείγματα εδώ στην Ευρώπη όπου προβλέπονται μέτρα της ε, κοινότητας, για παράδειγμα, για την κράτηση, αλλά και στο Μεξικό και τον ε, Παναμά απαγορεύεται η κράτηση μεταναστών. Να σας δώσω ένα πολύ καλό παράδειγμα από μια χώρα που δεν θα το περιμένατε, τη Γεμένη, όπου υπάρχει ένα λακτικό σύστημα φροντίδας που βασίζεται σε σπίτια για μικρές ομάδες ε, που δημιουργήθηκε από την ύπατη αρμοστία ε, μαζί με ε, ανθρώπους από τον χώρο των προσφύγων. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να μην θεωρείτε οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε να αποτελούν δικαιολογία για να μην ε, τηρήσετε τα δικαιώματα των παιδιών και της ερήτρες της σύμβασης. Ξέρω πολύ καλά ότι η κύρωση της σύμβασης για τα άτομα με αναπηρία αποτέλεσε πολύ σημαντικό βήμα, αλλά ε, όσον αφορά την σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, τα κράτη-μέλη μπορούν να ξεκινήσουν την όλη συζήτηση. Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ε, σύμβαση, ώστε να τεθεί η σύμβαση αυτή σε πολύ πιο ισχυρό πλαίσιο. Όσον αφορά τον καθορισμό της ηλικία, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου ε, γίνεται κατάχρηση του θέματος της ηλικία. Κανένας σόφρονος άνθρωπος δεν θα υποστήριζε την κατάχρηση της διαδικασίας, διότι αυτή υπονομεύει τα δικαιώματα και τις ε, ευκαιρίες για τα παιδιά ε, που ε, δικαιούνται να υποφεληθούν από το σύστημα. Ως Επιτροπή, λοιπόν, λέμε ότι οι μέθοδοι καθορισμού της ηλικίας που βασίζονται μεταξύ άλλων στην ανάλυση των οστέων θα πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά και ιδιαίτερα για παιδιά ηλικίας 16 έως 18 ετών αναγνωρίζουμε ότι οι, μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ε, για τον καθορισμό της ηλικία ε, είναι ε, λυπής σε πολλές περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν διατομεακές εξετάσεις όπου να συμμετέχουν και ψυχολόγοι, για παράδειγμα, και άλλοι. Εάν γίνεται αποκλειστικά γιατρική εξέταση, αυτή θα πρέπει να είναι ε, μη παρεμβατική. Ε, υπάρχουν παιδιά που δεν θέλουν να περάσουν από αυτή τη διαδικασία και θέλουν ότι δεν πειράζει, ενήλικας είμαι. Επίσης, όσον αφορά τα παιδιά που εξαφανίζονται, δεν ξέρω... Ε, αν τα στοιχεία που έχετε όντως ε, είναι επιβεβαιωμένα. Εγώ έχω ακούσει για 10.000, αλλά θα πρέπει να ε, εξετάσουμε το ρόλο που θα πρέπει να παίξουν ε, οι αξιωματικοί επιβολές του νόμου. Διότι τα παιδιά που εξαφανίζονται σημαίνει ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας. Θα πρέπει οι αρχές επιβολής του νόμου να φροντίζουν να μην εξαφανίζονται παιδιά. Επίσης υπάρχει έλλειψη διαδικασιών για την ε, κυδαιμονία. Τα παιδιά αυτά ε, στα κέντρα υποδοχής ε, συχνά έχουν πολύ κακές συνθήκες υγιεινής και υφίστανται βία. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τα παιδιά αυτά να πούν τις απόψεις τους και να, να κάνουν παράπονα σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Σε κάποιους από αυτούς τους καταβλισμούς τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν ντους, δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα ε, και υπάρχουν περιπτώσεις όπου κακοποιούνται από ενήλικες. Ε, ε, είχαμε περιστατικά όπου τα παιδιά πρέπει να πληρώσουν για να έχουν πρόσβαση στους καταβλισμούς. Και όλα αυτά φυσικά ε, δεν αποτελούν συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά την ε, επανένωση οικογενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετές από τις συστάσεις μας Μάλλον θα σας παρουσιάσω κάποιες από τις συστάσεις μας. Ε, η σύμβαση δεν ε, απαγορεύει τον χωρισμό της οικογένειας, αλλά λέει ότι δεν ε, θα πρέπει να γίνεται αυτό ενάντια στη θέλησή τους, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές θεωρήσουν ότι αυτό είναι προς συμφέρον του παιδιού. Μπορεί λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του παιδιού να υπαγορεύει ε, αποχωρισμό από την οικογένεια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται διοικητική αλλά και δικαστική εξέταση και ότι θα πρέπει να ε, συμμορφωνόμαστε με τα κριτήρια περί ε, συμφέροντος του παιδιού. Και όσον αφορά την επανένωση της οικογένειας, εδώ μας ενδιαφέρει ο ορισμός της οικογένειας. Θα πρέπει επίσης ο καθορισμός αυτός να γίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα. περιπτώσεις όπου η διαδικασία και η σε δεν γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση. Για παράδειγμα, ε, διαρκούν πάρα πολύ ή υπάρχει ένας άνθρωπος ε, αρμόδιος ε, για 50-60, έχω ακούσει και για εκατοντάδες παιδιών. Πώς μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε την σωστή κυδαιμονία τη στιγμή που είναι κανείς αρμόδιος για πάρα πολλά παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αμεροληψία στη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει να ακούμε τα παιδιά, θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, θα πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμέ ε, για να διαπιστωθούν οι οικογενειακοί δεσμοί. Και όλα αυτά θα πρέπει να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία. Επίσης, ε, ε, κατάρτιση για τους κυδεμόνε και επαρκής οικονομική και ανθρώπινη πόρη. Ε, με ρωτήσατε τι εννοούσα όταν μιλούσα για κατάρτιση, μιλούσατε για ε, χρήση νέων επαγγελματιών. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Υπάρχει εντύπωση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι απαραίτητοι επαγγελματίε, ε, κοινωνική λειτουργοί, ε, κυδεμόνε, κοινωνιολόγοι κλπ. βρίσκονται σε θέση να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Εμείς ως Επιτροπή απαντάμε όχι, ακόμα και αν υπάρχουν το επίπεδο των γνώσεών τους για τα δικαιώματα του παιδιού είναι πολύ περιορισμένο. Ε, και αυτό ξεκινάει από αυτούς ε, που ε, συμμετέχουν στις αποστολές της Frontex. Τα εγχειρίδια κατάρτισής τους μιλούν για τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά πώς διασφαλίζεται αυτό. Θα πρέπει λοιπόν όσοι εργάζονται με τα παιδιά να έχουν ε, τα απαραίτητα προσόντα. Και συχνά ξεχνάμε και την ε, ψυχολογική βία που υφίστανται τα παιδιά. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν έχουμε τους απαραίτητους ανθρώπους, το απαραίτητο προσωπικό για να παράσουμε σωστές υπηρεσίες στα παιδιά αυτά. Και κλείνω σιγά σιγά. Τέθηκε και το θέμα της εμπορίας ανθρώπων, ε, τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να σας δώσω νούμερα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές. Ε, σημείο κίνησης είναι πάλι η νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές. Είδαμε χώρες ε, με πολύ χαμηλές ε, ποινές. Θα πρέπει να αλλάξει η δυναμική. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν σε δραστηριότητες εμπορίες, εμπορίας γυναικών. Η ιδέα λοιπόν ότι ε, ότι ε, ένας ε, υπέρβαρος άντρας με κινητό στο, με κινητό στο κάθε χέρι κλπ. είναι αρμόδιος για κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητα η σωστή εικόνα. Και ένα στοιχείο που προκύπτει είναι ότι δεν είναι θέμα το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εντός σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ένα θέμα οριζόντιο στην Αφρική, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική. Κάποιες χώρες είναι χώρες ε, διέλευσης, ε, κάποιες είναι χώρες προέλευσης, ε, κάποιες χώρες είναι χώρες προορισμού, κάποιες χώρες είναι συνδυασμό όλων αυτών. Οι χώρε όπου έχει σημειωθεί πρόοδο, η Μπουρκίνα Φάσο, η Γουινέα κλπ. είναι αυτέ που υπέγραψαν μνημόνιο κατανόηση και δημιούργησαν ειδικέ ομάδε εντό των διαφόρων υπουργείων για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει τη εμπορία ανθρώπων. Μία παρατήρηση ακόμα και θα κλείσω. Ήδη μίλησα για τον καθορισμό της ηλικίας και θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που έθιξε ε, ο φίλανδος Ευρωβουλευτής. Πράγματι υπάρχει κατάρτιση, κατάχρηση όσον αφορά τον καθορισμό της ηλικία, αλλά είναι σημαντικό για τα κράτη και το είδαμε αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα όπου η ε, ε, εφημερίδε στο Ηνωμένο Βασίλειο είπαν ότι τα παιδιά που βγήκαν από το καλέ φαίνονται πολύ μεγαλύτερα και ε, κάνουν κατάχρηση του συστήματο. Αλλά οι υποχρεώσεις μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να αποτελούν παιχνίδι για, για τον τύπο. Δεν θα πρέπει ο τύπος να μας κάνει να ξεφύγουμε από τις υποχρεώσεις μας. Ε, και μια τελευταία παρατήρηση, ξέρω ότι με πιέζει ο χρόνος. Ως Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού προσπαθούμε, μάλλον συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Εάν όμως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού τεθεί στο επίκεντρο των εργασιών σας, εάν ε, έχετε μελέτη αντικτύπου στα δικαιώματα του παιδιού στις πολιτικές σας, εάν το συμφέρον του παιδιού αποτελεί το κριτήριο και για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές σας δράσεις, τότε πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης. Και εάν υπάρχει τρόπος να στηρίξουμε τη διαδικασία αυτή, θα χαρούμε πολύ. Ένας από τους συναδέλφους που συμμετέχει στην εκπόνηση της ε, σχετικής οδηγίας. είναι γνωστό μου και αν μπορέσει η Επιτροπή της, ε, για τα Δικαιώματα του Παιδιού να συμμετάσχει, να συμβάλλει στη διαδικασία, ε, θα το κάνουμε πολύ ευχαρίστως. Και τόσα χρόνια μετά την ε, υπογραφή της ε, σύμβασης, ε, το συμφέρον του παιδιού αποτελεί ακόμα το γνώμονα για καλές λύσεις με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ε, ήταν πρόταση της Επιτροπής μας να σας προσκαλέσουμε, ήταν επιθυμία της Επιτροπής μας να σας προσκαλέσουμε για να ενημερωθούμε για το έργο σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που δεχτήκατε την πρόσκληση που μας ε, συζητήσατε μαζί μας όλα αυτά τα θέματα, τα θέματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Ε, Από τη συζήτηση φαίνεται επίσης από το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, για παράδειγμα για τις διαδικαστικές εγγύσεις στις ανήλικους ποινικές διαδικασίες και από άλλα θέματα, φαίνεται πόσο μεγάλος, μεγάλη σημασία αποδίδουμε στα δικαιώματα του παιδιού. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ο θα αναλάβει την Προεδρία τη Επιτροπή μα για το επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη. Thank you very much, Claude. Ευχαριστώ πολύ, Claude. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Πρόκειται για μια μελέτη για τον κυβερνό εκφοβισμό νεαρών ε, ε, η οποία ζητήθηκε από την ε, Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ζητήθηκε να εκπονηθεί αυτή η μελέτη γιατί πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο εξαπλώνεται οργά και απειλεί ανήλικους, νέους. Η Επιτροπή δημοσιοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2014 και ε, αναφέρεται σε στην κατάσταση του προβλήματος, κάνει έναν απολογισμό της κατάστασης, ε, αναφέρει ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, πώς θα πρέπει να αναλυφθεί ε, δράση σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα για παράδειγμα στον τομέα της ε, εφαρμογής 2011-93 για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θα δώσω τον ε, λόγο στην ε, κυρία Ντάλα Πότσα, η οποία ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση της μελέτης, για να μας την παρουσιάσει. Κυρία Ντάλα Πότσα. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να καταγραφούν οι μορφές και οι τρόποι με τους οποίους ασκείται ο κύβερνο εκφοβισμός ε, σε όλα τα 28 κράτη-μέλη ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας ακόμα περισσότερο σε 9 κράτη-μέλη για μεγαλύτερη ανάλυση της κατάστασης εκεί. Αναφερόμαστε σε νέους κάτω των 18 ετών. Η μεθοδολογία συμπεριλαμβάνει συνδέξεις με νέους και ενδιαφερόμενους. Αυτή τη στιγμή ούτε σε διεθνές ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ένας ε, συγκεκριμένος ε, και κοινά αποδεκτός ορισμός του κυβερνοευκφοβισμού. Ε, Μόνο λίγα κρατημέλη έχουν υιοθετήσει έναν τέτοιον ορισμό. Και υπάρχει μεγάλη, μεγάλη ποικιλομορφία, μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους ορισμούς που έχουν δοθεί. Ωστόσο υπάρχει συμφωνία ως προς το ότι ο κύβερνοεκφοβισμός είναι μια πρακτική βίαιης, ε, βίαιου εκφοβισμού, απειλή ενάντια ενό ανθρώπου που δεν έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί ο ίδιο και η οποία πρακτική συχνά επαναλαμβάνεται. Έχει ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά. Ε, ο κυβερνοεκφοβισμός είναι ε, μια πρακτική την οποία γίνεται μέσω των μέσων των ηλεκτρονικών. Εδώ υπάρχει μια αναντιστοιχεία ανάμεσα στην ε, ισχύ που έχει ο φίτης και το θύμα. Ο φίτης έχει τη δυνατότητα να παραμείνει ανώνυμος και εκμεταλλεύεται αυτή τη δυνατότητα. Συχνά ο κυβερνοεκφοβισμός γίνεται με τέτοιον τρόπο που δημοσιοποιείται και γίνεται γνωστός ε, και ε, σε χιλιάδες άτομα έχει αναφερθεί αύξηση των περιστατικών κυβερνοεκφοβισμού στα παιδιά από 11 έως 16 ε, ετών από 7% στο 12%, το 12% το 2014, δηλαδή σε μια περίοδο ε, τριών ετών, τεσσάρων ετών. Ε, βέβαια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, για αυτά τα στοιχεία γιατί ε, όπως σα είπα οι ορισμοί που δίνονται από τη μία χώρα στην άλλη είναι διαφορετικοί. Πολύ συχνά υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στου ορισμούς που χρησιμοποιούν κάθε, κάθε μελέτη. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες γενικές τάσεις που μπορούμε να εντοπίσουμε. Για παράδειγμα, είναι πιο πιθανό τα θύματα να είναι θύτες ε, παρά να μην τους έχει αγγίξει το θέμα. Επίσης, στον στις περιπτώσεις κυβερνοεκφοβισμού ε, συχνά ε, διαπιστώνουμε ότι το θύμα μπορεί να έχει υποστεί και άλλου τύπου εκφοβισμό, ε, άλλου είδους bullying πιο νωρίς. Επίσης διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση όσον αφορά το φύλλο του θύματος. Υπάρχει μια, είναι ένα φαινόμενο, ένα πρόβλημα που αγγίζει και τα κορίτσια και τα αγόρια εξίσου. Επίσης δεν υπάρχει ένα κοινό νομικό ε, πλαίσιο που να, για την καταπολέμηση του εκφωνισμού. Ωστόσο, συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 ε, και 31 της ε, Σύμβασης του ΟΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Υπάρχουν ορισμένα ε, πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που η ε, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα ή επίσης η Σύμβαση για, το, την Καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που μπορούν να αξιοποιηθούν για την καταπολέμηση του, του κυβερνοεκφοβισμού. Από την πλευρά του ΟΗΕ έχει καταρτήσει ένα ε, πλαίσιο πολιτικής το 2014 με ένα ψήφισμα για την προστασία των παιδιών από τον κυβερνοεκφοβισμό. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης έχει υιοθετήσει μια στρατηγική που θέτει την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ε, στο ίντερνετ ε, ως μία από τις προτεραιότητές της για την περίοδο 2016-2021. <clears throat> Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, εδώ έχει μόνο ε, υποστηρικτικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της. Ωστόσο, έχουν υιοθετηθεί ε, οδηγίε συναφή με το θέμα, όπω για παράδειγμα η οδηγία για την καταπολέμηση τη ε, ε παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών ή η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Αυτά συνδέονται με το ζήτημα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει μια, ένα συγκεκριμένο, μια ξεχωριστή νομοθεσία για το ζήτημα. Στη, κατά την 25η επέτειο της ε, Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ε, ψήφισμα στις 27 Νοεμβρίου του 2014, στο οποίο αναφερόταν και η ανάγκη της καταπολέμησης του κυβερνοεκφοβισμού. Η καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών και online συμπεριλαμβάνεται στο λόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού. Έχει επίσης υιοθετήσει μια σειρά πολιτικών η Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, την ε, βελτίωση της ασφάλειας online. Όπως για παράδειγμα τη στρατηγική του 2012 της Κομισιόν τη Επιτροπής για ένα καλύτερο ίντερνετ για τα παιδιά. Έχει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προγράμματα οικονομικής βοήθειας για τη δημιουργία συστημάτων προστασίας των παιδιών στο εθνικό επίπεδο. Ε, κανένα από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ένα, μια ξεχωριστή νομοθεσία, μια νομοθεσία επικεντρωμένη ειδικά στο ζήτημα του κύβερνου εκφοβισμού. Ωστόσο, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν το θέμα στο πλαίσιο άλλων ποινικών δικημάτων, όπως για παράδειγμα της απειλής, της βίας, της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 14 ε, κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές για το θέμα ή για συναφή θέματα, όπως για παράδειγμα την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, την ενημέρωση για τα θέματα αυτό στα σχολεία, την προστασία του παιδιού στη, ε, online έχουμε ε, διαπιστώσει ε, βέλτιστες πρακτικές σε μια σειρά Ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Εστονία, η Γερμανία, 100 χώρες, η Ιταλία ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και άλλες. Δηλαδή, πρακτικές οι οποίες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση του φαινομένου του εκείβερνου εκβοβισμού και στην προστασία των θυμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε πρωτοβουλίες από το συνήγορο του παιδιού στην Ελλάδα και στην Εστονία. Έχουμε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά στη Γερμανία και στις κάτω χώρες ή ε, την ε, εισαγωγή προγραμμάτων εκπαιδευτικών στα σχολεία ε, προληπτικών και για, και για την καταπολέμηση του bullying. Μια άλλη βέλτιστη πρακτική, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η συμμετοχή των ιδίων των παιδιών στην εκπόνηση των πολιτικών που τα αφορούν. Στι κάτω χώρε υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά για να μάθουν ε, την αξία του σεβασμού του άλλου και. Μια άλλη βέλτιστη πρακτική ήταν ε, η δημιουργία ειδικών ε, δυνατοτήτων στις σελίδες έτσι ώστε κάποιο να μπορεί άμεσα να καταγγείλει ε, μια ε, σελίδα η οποία, μέσω της οποίας γίνεται εκφοβισμό. και επίσης μια άλλη βελτιστή πρακτική που διαπιστώσαμε είναι η δημιουργία ειδικών δομών για την υποστήριξη των θυμάτων στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Οι συστάσεις μας Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να, υιοθετήσει σε, να, να, αναλάβει πρωτοβουλία έτσι ώστε να υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας ορισμός του εγκλήματος του κύβερνο-εκφοβισμού. Αυτό θα βοηθήσει στην εναρμόνιση ε, και θα βοηθήσει όλα τα κράτη να ξεφύγουμε από την σημερινή κατάσταση όπου κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του ορισμό. Θα ήταν επίσης ευχής έργων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την ε, ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών αλλά επίσης και με την εμπλοκή του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα εκείνων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαδικτύου και ακόμα περισσότερο στον τομέα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και εκείνο ένα ρόλο να παίξει, διασφαλίζοντα ότι το, ο κυβερνοεκφοβισμό παραμένει υψηλά στην ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα τη ε, συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί τις που αναλαμβάνει η Επιτροπή στον τομέα αυτό ε, για να εξασφαλίζει ότι το ζήτημα του κυβερνοϊκορισμού δεν θα ξεχνιέται, δεν θα ε, παραλείπεται ε, στην χάραξη πολιτικής. <clears throat> Χρειάζεται επίσης να να ε, μεγαλύτερη, να, να προωθηθεί ένας μεγαλύτερος ρόλος, σημαντικότερος για το συνήγορο του παιδιού. και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες, τις δεξιότητες στον τομέα του χειρισμού του διαδικτύου και για τα παιδιά και για τους γονείς τους. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τελαπότσα και να ξεκινήσει τώρα ο ε, γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων. Δεν ξέρω, συνάδελφοι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Η κυρία Κινίτσι. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή της πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ε, και ε, την ευάθυνση στον εκφοβισμό μεταξύ των νέων. Είναι ένα θέμα δυστυχώ ε, το οποίο ε, διαιωνίζεται και είχε και τραγικές συνέπειες, διότι πολλοί νέα παιδιά, θύματα του κυβερνοεκφοβισμού, ε, έχουν προβεί και σε ακραίες ε, πράξεις. Επομένως και ως συμπρόεδρος της ομάδος για τα δικαιώματα των ανηλίκων θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε τη μέγιστη προσοχή στο θέμα αυτό. Σήμερα παρουσιάστηκαν μία σειρά από πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες σκέψεις, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ και να ρωτήσω ε, την ε, προσκεκλημένη μας εάν ε, μπορούμε να εξετάσουμε κάτι υπό ένα διπλό προφίλ. Καταρχάς το προφίλ της πρόληψης, διότι πέραν των νομοθετικών λύσεων που θα μπορούσαν να δοθούν και πρέπει να δοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών και η χώρα μου η Ιταλία προχωρά κάποια ε, πράγματα και θέλει να έχει πολύ σύντομα νομοθεσία για τον κυβερνοεκφοβισμό. Πέραν όμως ε, των νομοθετικών παρεμβάσεων είναι πάρα πολύ σημαντική η πτυχή της πρόληψης κατ' εμέ. Η πρόληψη η οποία θα πρέπει ε, σίγουρα να ανατίθεται στα σχολεία αλλά και στην οικογένεια. Αλλά δεν είναι πάντα σε θέση οι γονείς ε, να βοηθήσουν τα παιδιά τους ε, να χρησιμοποιούν ε, με συνειδητό τρόπο τα μέσα της πληροφορικής επιστήμης. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψή σας επ' αυτού πώς μπορούμε να έχουμε πρόληψη η οποία να είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και η άλλη πτυχή, την αναφέρατε κι εσείς, είναι η πτυχή της ε, στήριξης και της προστασίας ε, ε, του κυβερνοεκφοβισμού. Γνωρίζουμε ότι ο εκφοβισμός είναι μια μορφή δίωξης με απλούς όρους για κάποιον πιο αδύναμο, κάποιον τον οποίο εντοπίζουν κάποιοι ως πιο αδύναμο, τον οποίο διώκουν και καταδιώκουν ορισμένες φορές και μέσω ε, της πληροφορικής αυτή τη στιγμή και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να υποστηρίξουμε καταλήλως τα θύματα αυτής της μορφής συμπεριφορών. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει καταγγελία για ε, κάποιον ότι είναι θύμα εκφοβισμού ή ε, κύβερνο εκφοβισμού. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον λοιπόν ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την ε, κατάσταση για να μπορέσει να σταματήσουν αυτές οι ακραίες συμπεριφορές. Ε, υπάρχει για παράδειγμα παράδειγμα η περίπτωση ενός κοριτσιού που λεγόταν Καρολίνα στην Ιταλία 14 ετών η οποία αυτοκτόνησε γιατί ήταν θύμα εκφοβισμού μέσω Facebook. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ε, για πρόληψη εφενός και ταυτόχρονα και για κατάλληλη στήριξη στα θύματα ε, περιπτώσεων εκφοβισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπιθ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένες φορές εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχουμε μια ακρόαση που είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι συζητούμε ανεπίσημα για θέματα τα οποία ε, αξίζουν ε, τον κόπο να τα συζητήσουμε, να προβληματιστούμε. Ε, τι ε, προτείνουμε και ε, για να, κάποια θέματα για τα οποία αξίζει να δώσουμε έναν αγώνα. Αλλά μας λείπουν κάποια στοιχεία ορισμένες φορές. Κάποιες λοιπόν από αυτές τις ακρόσεις μας παρέχουν αυτά τα εργαλεία και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη διεξοδική παρουσίαση. Με κανάντα να σκεφτώ και τις συνέπειες του κυβερνοεκφοβισμού και τον τρόπο με τον οποίο ε, μάθαμε για αυτό το φαινόμενο και ίσως ε, θα μπορούσατε να μας αναπτύξετε λίγο περαιτέρω το θέμα, ώστε να έχουμε κάποια περαιτέρω στοιχεία. Το πρώτο θέμα είναι ε, τι φέρπει ε, πίσω από τον κυβερνό εκφοβισμό. Πρόκειται για κάτι από ό,τι φαίνεται που είναι ένα περίπτωση διαφορετικό φαινόμενο. Προφανώς, έτσι φαίνεται, αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι παραπάνω. Μπορεί να υπάρχει κάποια μορφή οργανωμένου εγκλήματος, η οποία να ανακύπτει ε, και να προκύψει ίσως μελλοντικά στον ορίζοντα. Είναι σε επαφή μεταξύ τους ε, αυτοί οι άνθρωποι που ε, εκφοβίζουν άλλους, είναι οργανωμένοι με κάποιο τρόπο, ανταλλάζουν εμπειρίες, εμπορεύονται με προϊόν ε, την πίεση ή τον εκφοβισμό ε, έναντι ανυπεράσπιστων ε, νέων αγοριών και κοριτσιών ή παιδιών. Και το άλλο αφορά την ισορροπία που πρέπει να εξευρεθεί μεταξύ της αντίληψης ότι ο κυβερνοεκφοβισμός είναι στην πραγματικότητα μια απειλή για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των νεότερων και τη σημασία του να γίνεται σεβαστή η αυτονομία αλλά και η ιδιωτική ζωή των νέων ανθρώπων. Διότι και βάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν δικαίωμα στην ιδιωτική του ζωή. Εξ όσων γνωρίζουμε, πολλές περιπτώσεις κυβερνοεκφωνισμού διαπιστώνονται από τους γονείς επειδή ψάχνουν τι κάνουν στο διαδίκτυο τα παιδιά τους ή οι νεότεροι, ε, τα νεότερα μέλη της οικογένειας και με παράνομο τρόπο, διότι πρέπει να παραβιάσουν και την ιδιωτική ζωή των νέων παιδιών για να μπορέσουν να μάθουν. Πρέπει κάπως να παρέμβουν και επομένω ε, ψάχνουν τα τηλέφωνά τους, τα τάμπλετ τους, τους προσωπικούς τους υπολογιστές, ορισμένες φορές είναι υποχρεωμένοι για να μάθουν τι συμβαίνει. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια παραπάνω από αυτού. Ευχαριστώ. Ωραία, να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Ντελαπότσα για να απαντήσει στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις και να ε, έχετε κατά νου ότι έχουμε καθυστερήσει λίγο. Επομένως αυτή απλώς θα είναι μια αρχή μια συζήτησης, αλλά να ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις σας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση και την ε, ε, προσέγγιση της πρόληψης τα ευρήματα της μελέτης μας ε, υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, εκπαίδευση που είναι ο βασικός παράγων επιτυχίας ε, στην πρόληψη. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα εκπαίδευσης σε επίπεδο κρατών μελών που είναι αποτελεσματικά στη μείωση του κυβερνοεκφοβισμού. Για παράδειγμα το πρόγραμμα ΚΙΦΑ το οποίο ξεκίνησε στη Φιλανδία και μετά εφαρμόστηκε και σε διάφορες χώρες και στις κατοχώρες και το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση για το σχολείο και περιλαμβάνει όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας και στο σχολείο και να συμμετέχουν τα παιδιά στην εξέβρεση λύσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό ε, παράδειγμα ενός προγράμματος το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Όσον αφορά τη στήριξη προ τα θύματα, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, τα πορίσματα της μελέτης ε, για ε, τα νέα παιδιά για ηλικίες 12 έως 21 ετών ε, μας υποδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρχει υποστήριξη των σημάτων, κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι τα παιδιά θέλουν επίσης ε, ε, να τους υποστηρίξουν όσο αφορά τη δίωξη των δραστών και να μπορέσουν οι δράστες να καταλάβουν ε, και τι συνέπειες έχει η συμπεριφορά τους και να αντιληφθούν τι σημαίνει να βρεθούν στη θέση του θύματος. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την ερώτησή σας. Όσον αφορά ε, την πτυχή του κυβερνοεγκλήματος, ο κυβερνοεκφοβισμός είναι αναγνωρισμένη μορφή κυβερνοεγκλήματος. Είναι πολύ επικίνδυνο ούτως ή άλλως και σύμφωνα με μία έρευνα ένα εκατομμύριο θύματα κυβερνοεγκλήματος περιλαμβάνουν και θύματα κυβερνοεκφοβισμού. Άρα το κύβερνο ο κυβερνοεκφοβισμός είναι μία μορφή κυβερνοεγκλήματος. Όσον αφορά την ε, δέουσα ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή των παιδιών και την παρέμβαση των γονέων τους, ε, και εδώ να τονίσω ότι η έρευνα μεταξύ των νέων ανθρώπων ε, που διεξάγαμε κατέδειξε ότι τα παιδιά επισημαίνουν ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος γονικός έλεγχος και έλεγχος από πλευράς εκπαιδευτικών ε, για τη συμπεριφορά του στο διαδίκτυο. Από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά θα ήθελαν οι γονείς και οι ε, εκπαιδευτικοί να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι και να έχουν καλύτερες δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να, σκα... τους κατευθύνουν για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη μελέτη σας. Η μελέτη είναι διαθέσιμη, επομένως ε, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως περαιτέρω τροφή για σκέψη. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη τώρα. Η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις συνέπειες των ε, ε, big data. Ε, η συγγήτρια είναι η κυρία Αναγκόμε, η οποία θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση της τώρα. Ε, σας διανεμήθηκε στις 27 Οκτωβρίου το έγγραφο. Η Αναγκόμε λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, είπατε και εσείς, ε, έχουν οι συνάδελφοι την έκθεση μπροστά τους. λόγω των περιορισμών ε, το έγγραφο αυτό αποτελεί περίληψη των όσων θα έπρεπε να περιέχει. Ε, αλλά περιμένω να δω τις τροπολογίες των συναδέρφων, θα υποβάλω και εγώ κάποιες για να αναπτύξουμε κάποιες από τις βασικές ιδέες που περιέχονται στο έγγραφο. Τρεις βασικούς τομείς ε, αφορά η έκθεση αξιολόγηση της κατάστασης, ε, αντίκτυπος ε, των ε, μαζικών δεδομένων στη χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς και τρίτον για σκοπούς επιβολής του νόμου. Βέβαια, κάποιες από τις ανησυχίες μας αφορούν και, αφορούν και τους τρεις αυτούς τομείς. Όπως είπα, είχαμε περιορισμούς όσον αφορά ε, την έκταση του εγγράφου. Οι τροπολογίε όμω μπορεί να μα βοηθήσουν να συμπεριλάβουμε πράγματα που δεν συμπεριλαμβάνονται ή που συμπεριλαμβάνονται δεν τονίζονται όμω επαρκώ. Αναγνωρίζουμε ότι οι εξελίξει ε, στην τεχνολογία και ότι ε, η γενική χρήση ε, ηλεκτρονικών συσκευών έχουν προσφέρει ευκαιρίες σε επιχειρήσεις, πολίτες και κυβερνήσεις ενέχουν όμως και σημαντικούς κινδύνους όσον αφορά την προστασία των θεμελιωτών δικαιωμάτων, ε, της ιδιωτικής ζωής ε, και την αποφυγή των διακρίσεων. Επίσης, ε, το να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση μασικά δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα με ε, επιβλαβή συνέπειες για τους πολίτες. Τον Μάιο είχαμε επισκεφτεί την Silicon Valley και μας είπε ένας από τους συνομιλητές μας ότι τα μαζικά δεδομένα ουσιαστικά είναι στατιστικές ε, που μεγεθύνονται με χρήση ενός αλγόριθμου. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό, δεν νομίζω όμως ότι ε, αποτελεί σωστή περιγραφή της πραγματικότητας. Ε, κάθε στατιστική όμως μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χειραγώγησης ε, και αν χρησιμοποιεί κανείς μέσα για να μεγεθύνει και όλες τις στατιστικές αυτές, ε, τότε και οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. και μας ενδιαφέρουν βέβαια ιδιαίτερα οι επιπτώσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, η μη διάκριση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και οι συνομιλητές μας ε, ανέφεραν ε, τις συνέπειες για παράδειγμα στον τομέα των ασφαλίσεων. ή, ε, την, τον τομέα, ή στον τομέα της υγείας. Ε, είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει εμπιστοσύνη του κοινού ε, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με σωστή επιβολή του νόμου. Δεν προτείνουμε νέα νομοθεσία με την έκθεση αυτή. Έχουμε την εφαρμογή του, της δέσμης μέτρων που υιοθετήθηκε ε, υπό τη δική σας καθοδήγηση κύριε Πρόεδρε και το σημαντικό είναι πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις αρχές ε, προστασίας δεδομένων και το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Πιστεύω ότι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η λογοδοσία είναι σημαντικές αξίες και ότι είναι οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν ε, την ε, εφαρμογή. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην περίπτωση των ε, βάσεων δεδομένων που έχουν μεγάλες επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν δεδομένα για, για μεμονωμένα άτομα τα οποία τα πολλούν και σε άλλους, τα διαβιβάζουν σε υπεργολάβους κλπ. η ενίσχυση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ε, προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Δεν νομίζω όμως ότι το αναγνωρίζουν αυτό όλοι. Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι και μάλλον ε, κανείς δεν συνειδητοποιεί την διάσταση των κινδύνων αυτών. Επιμένω ότι χρειαζόμαστε πλατφόρμες ε, διαλόγου ανάμεσα σε δημόσιες αρχές ε, και ιδιωτικούς φορείς. Τις επιχειρήσεις δηλαδή που ε, έχουν βάσεις δεδομένων, με μαζικά δεδομένα και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτών των ε, αλγορίθμων. Ζούμε σε έναν κόσμο ε, δικτύων, ε, εφαρμογών του διαδικτύου. Και η χρήση των διαφόρων προϊόντων δεν σημαίνει απαραίτητα η ικανοποίηση του καταναλωτή με τα προϊόντα αυτά, αλλά μπορεί απλά να ε, δείχνουν την ε, απογοήτευσή τους ε, και το ότι συμβιβάζονται με τα προϊόντα που μπορούν να βρουν. Ζούμε πια στον κόσμο του ίντερνετ των πραγμάτων. οι τράπεζες, ε, η αεροπορία, ε, πολλά συστήματα βασίζονται στην αξιοπιστία των βάσεων δεδομένων, ε, κάτι που επίσης βασίζεται στην συμμόρφωση με, τον, το δίκαιο περί δικαιωμάτων. Αυτά έχω να πω για τη συζήτηση αυτή. Περιμένω να ακούσω ε, τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και να δω τις τροπολογίες τους για να συμβάλλουν στη βελτίωση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρει ευρωβουλευτέ και εγώ ίδιο θα θέλω να πάρω το λόγο. Πρώτα το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Άννα ε, για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Θετικό βρίσκω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί καλή βάση για συζήτηση. Κατά τη γνώμη όμως ε, δεν ε, είναι επαρκής όσον αφορά το τι μπορεί, μπορούν να πετύχουν τα μαζικά δεδομένα και πώς επηρεάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί η έκθεση αυτή. Υπάρχει εδώ και η προσπάθεια να οριστούν τα μαζικά δεδομένα και να περιγραφούν τα πλεονεκτήματά τους ε, αυτό το βρίσκω καλό, διότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε πια τα μας δεδομένα, αποτελούν πραγματικότητα και τα έχουμε στις κοινωνίες μας. Ε, το ε, θέμα είναι πώς θα τα χειριστούμε. Στο ε, ε αναφέρεται η ευρεία χρήση των αισθητήρων για συγκέντρωση δεδομένων. Αναρωτιέμαι λοιπόν, πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα θεμελιώδη δικαιώματα ή πρόκειται για ανωνυμοποιημένα δεδομένα με τα οποία δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε εις βάθος. Επίσης, οι αλγόριθμοι θα πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω και θα πρέπει να φροντίσουμε να παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα των δεδομένων και να μην οδηγεί σε λάθος αποφάσεις. Όσον αφορά την ανασφάλεια των πολιτών, εγώ τη βλέπω κάπως διαφορετικά. Οι πολίτες σε βλέπουν τι τους φέρνει το μέλλον Γνωρίζουν βέβαια ότι στον τομέα των δεδομένων έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Ο όρος μαζικά δεδομένα μπορεί να οδηγεί σε ανασφάλεια, αλλά ε, αυτά καθ' αυτά τα, βασικά, τα μαζικά δεδομένα δεν θα πρέπει να οδηγούν σε ανασφάλεια, διότι, για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας μπορεί να γίνει σωστή η χρήση τους ε, και να πετύχει κανείς πολλά για την ε, καλύτερη καταπολέμηση των ασθενειών, ε, για την καλύτερη χορήγηση φαρμάκων. Πράγματα που μπορεί να πετύχει κανείς με τη χρήση μαζικών δεδομένων. Όσον αφορά τις τεχνικές ψευδονυμοποίησης ή εκειάνομνημοποίησης στο σημείο 3, των προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα ε, εμπίπτουν στην νομοθεσία περί προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων. Ε, και έχουμε συζητήσει το θέμα. Η ψευδονιμοποίηση των δεδομένων αποτελεί τρόπο βελτίωσης των δεδομένων αυτών ή ευκολότερης χρήσης τους. Κατά τη γνώμη μου, ναι, μπορεί να υπάρχουν όμως και άλλες τεχνικές τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Όταν μιλάμε για την ψευδονιμοποίηση τέτοιων δεδομένων, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πώς μπορεί να γίνει πάλι η ταυτοποίηση. Δεν είναι κακό το να έχουμε χρήση των μαζικών δεδομένων ε, εφόσον ε, έχουμε ψευδονομοποίηση, αλλά η εκ νέου ταυτοποίηση είναι ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρω ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα έχει τεθεί σε ισχύ ε, ο κανονισμός ε, για ε, την προστασία δεδομένων, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα χειριστούμε την σχετική οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μαριλάουστιν. Παρακαλώ. And I also uh, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τη δυνατότητα τώρα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση και ελπίζω αυτή η συζήτηση να μην γίνει με βιασύνη. Γιατί το θέμα είναι δύσκολο, είναι περίπλοκο και καινούριο. Και έχουμε την σχετική εμπειρία ότι με τη συζήτηση να γνωρίζουμε και προβλήματα που δεν τα είχαμε φανταστεί και τα ανακαλύπτουμε. Επομένως θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση σε βάθος για να αντιληφθούμε ακριβώς και ποιες είναι οι εξελίξεις στις διάφορους τομείς. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω από όλους όσους συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση να έχουν διαβάσει πολύ καλά πρώτα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Γιατί η πρόταση αυτή θα πρέπει να φροντίσουμε να μην προσπαθήσει να ξαναανακαλύψει τον τροχό, αλλά αντιθέτως να προσθέσει ένα επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα. Είναι κάτι που το θυμάμαι από προηγούμενες συζητήσεις, όταν είχαμε συζητήσει για το ζήτημα του profiling, ενώ στην πραγματικότητα τα ζητήματα αυτά είχαν υπηρεσμιστεί. Επομένως, μαζί με την Άννα μπορούμε να αναζητήσουμε το επόμενο βήμα. Ένα θέμα που κατά την άποψή μου δεν ε, αντιμετωπίστηκε πλήρως και σωστά στον κανονισμό είναι το γεγονό ότι με τα μαζικά δεδομένα, με τα πικτάτα έχουμε πλέον τη δυνατότητα οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων να χρησιμοποιηθεί σαν να ήταν προσωπικά δεδομένα. Δεν μιλούμε πλέον μόνο για την αντιμετώπιση του, με την ψευδονιμοποίηση ή με την ανενοποίηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε ένα σύνθελο δεδομένων που μα δείχνει τις μετακινήσεις όλων των ανθρώπων σε μια μεγάλη γεωγραφική περίοδο. Δεν είναι, περιοχή, δεν είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά μπορεί να μα δώσουν στοιχεία που δεν θα τα είχαμε διαφορετικά για τα άτομα αυτά. Επομένως, θα πρέπει να σταθούμε, κατά την άποψή μου, στη ρύθμιση τη χρήση αυτών των δεδομένων. Όχι μόνο ε, και όχι τόσο μάλλον στο ζήτημα της επεξεργασίας. Πώς θα διαπιστώσουμε, πώς θα ρυθμίσουμε εμείς νομοθετικά ποιος αλγόριθμος είναι καλός και ποιο είναι καλό, κακός. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε μια πορεία παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουμε τον τρόπο της, ε, ε, των φαρμάκων. Δεν κοιτάμε να δούμε αν μια ουσία είναι και ο τρόπο με τον οποίο την ανακαλύψαμε ήταν καλό ή κακό, αλλά συζητάμε εάν είναι επιβλαβή ή όχι για τον ανθρώπινο οργανισμό. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Εξετάζω την αιτιολογική ε, σκέψη F, σίγμα Βλέπω ότι υπάρχουν τρεις κύριες περιοχές τις οποίες θα πρέπει να σταθούμε. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει με ένα ζήτημα τεχνικό που είναι η ποιότητα των δεδομένων, επαγγελματικού χαρακτήρα αν θέλετε. Αλλά υπάρχουν και δύο ακόμα περιοχέ. Αμέσω μετά. Και σε αυτές τις άλλες δύο περιοχέ θα πρέπει να εφαρμόσουμε ηθικές αξίες και αρχές. Γιατί δεν μιλάμε πλέον για την επεξεργασία, μιλάμε για τη χρήση. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι που χρειαζόμαστε νέου κανόνε. Δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται ακόμα αυτοί οι κανόνε, γιατί έχουμε μπροστά μα μια καινούργια κατάσταση. Αυτό το δεύτερο λοιπόν η χρήση. Και το τρίτο είναι η νομική διατύπωση που θα ε, επιλέξουμε και πιθανώς και οι ποινές. Για παράδειγμα, θα ε, πηγαίναμε τόσο μακριά και θα επιλέγαμε, για παράδειγμα, την λύση του να απαγορευτεί στην νομοθεσία η χρήση συγκεκριμένων τεχνικών ανάλυση δεδομένων όταν τα δεδομένα αφορούν παιδιά, για παράδειγμα. Μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Και κάτι ακόμα που δυστυχώ δεν το βλέπω στο, στην, στο προσχέδιο είναι το ζήτημα τη εκπαίδευση. γιατί μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε για τη διαφάνεια, αλλά εάν τελικά δεν έχουμε στην διάθεσή μας όλοι οι πολίτες κάποιες βασικές γνώσεις, για παράδειγμα τι σημαίνει αλγόριθμος, τι σημαίνει συσχέτιση, στατιστική συσχέτιση. Ωραία συζητάμε τη διαφάνεια, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Επομένως, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την εκπαίδευση ως ένα βασικό εργαλείο που θα δώσει στα υποκείμενα της εξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων τη δυνατότητα να καταλαβαίνουν τι γίνεται. πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε και τη διάσταση της εκπαίδευσης. Και έρχομαι στο ζήτημα που αναφέρεται στις διεκτικές αρχές. Εδώ δυστυχώς θα έλεγα ότι το, το ζήτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είδα κάτι καινούριο σε σχέση με αυτά που προβλέπονται ήδη στο Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εδώ είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα χρειαστούμε την υπερογνωμοσύνη ειδικών. Για παράδειγμα, στον τομέα τη ε, κλασική ε, κλιματολογική έρευνα ε, από τη φύση του αυτός, αυτή, αυτός ο τομέα, είναι κάπως αχθρικό στη χρήση των μαζικών δεδομένων, των big data, γιατί πάντα υπήρχε η λογική ότι πρέπει να υπάρξει μια ερμηνεία της, του όποιου ευρήματος εγκληματολογικά. Ε, δεν έχουμε εμβαθύνει όσο θα έπρεπε στο ζήτημα της αξιοποίησης των big data από τις αδιοκτικές αρχές. στην συζήτηση για την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο, τώρα ξεκίνησε μια συζήτηση για το τι τελικά θα σημάνει το ότι όλοι οι πολίτες έχουν αυτές τις μικρές συσκευέ που συλλέγουν διαρκώς προσωπικά δεδομένα και στοιχεία για αυτούς. Και δεν βλέπω να αντικατοπτρίζονται αυτές τις συζητήσεις που είχαμε εκεί ακόμα στο προσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, παρόλη τη μικρή κριτική που έκανα, πιστεύω ότι το προσχέδιο της Άννα είναι πολύ καλή βάση συζήτηση. Ο πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Θα ζητήσω από του επόμενου ομιλητέ όμω να σεβαστούν το χρόνο ομιλία, να μην ξεπερνούν τα τρία λεπτά για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση. Ε, ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για τη δουλειά της. Να επισημάνω ότι μας είπε ήδη η κυρία Γκόμες ότι δεν μπορέσαμε να επενδύσουμε πάρα πολύ στο ε, σχέδιο του κειμένου. Επειδή υπάρχει το θέμα το οποίο συζητούμε όμως, θα πρέπει να προσδώσουμε καλύτερο περιεχόμενο στο κείμενο και να καλύψουμε τα κενά και να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε το κείμενο που έχει ήδη προτείνει. Το κείμενο, όπως ε, είπαν και άλλοι, αποτελεί πολύ καλή βάση για την ε, συζήτηση. τα πράγματα αλλάζουν με πολύ σημαντική ταχύτητα και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι τα big data, αλλά τα smart data, δηλαδή η ευφυής χρήση των στοιχείων και των στατιστικών. Κάτι το οποίο ε, θέτει μια άλλη σειρά από ερωτηματικά και έχει και μια σειρά από προκλήσεις ε, σε επίπεδο ιδιωτικής ζωής, ασφάλειας, ελευθερίας έκφρασης και νέων ευκαιριών. Ε, και πιστεύω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχει μια τεράστια πλειοψηφία υπέρ της υποδειγματικής προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει όμως να είναι και λίγο ισορροπημένα τα πράγματα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα και να αγκαιόμαστε ελευθερία, ασφάλεια, ιδιωτική ζωή και οικονομική ανάπτυξη. Όπως ε, πολύ σωστά είπε και η κυρία Γκόμες ήδη, δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τα εργαλεία τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα προστασίας δεδομένων. Θεωρώ επίσης ότι δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι όσον αφορά την ασφάλεια αλλά και όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων, ένα εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, όπως ε, της ε, ΙΖΑ αλλά και τα όσα έχει κάνει και ο Ευρωπαίος ε, Διαμεσολαβητής για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των εθνικών συνηγόρων του πολίτη και του προ, επόπτη προστασίας δεδομένων θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας πολύ σημαντικός ρόλος που περιλαμβάνει όλους εμάς και ε, όλους εκείνους που ε, ασχολήθηκαν με το θέμα της προστασίας της προσωπικής ζωής. Υπάρχει ε, θέμα όσον αφορά το κίνδυνο της κλοπής δεδομένων και του ρόλου των big data. Υπάρχουν ε, κάποιοι επικείμενοι κίνδυνοι σε αυτή την περίπτωση. Ε, κάποιες περιπτώσεις είναι πιο ε, απλές, κάποιες άλλοι ανησυχούν λίγο λιγότερο. Πρέπει λοιπόν να παρέμβουμε για να υπάρχει πιο ενιαία δράση από πλευράς των μελών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Τώρα όπως ο συνάδελφος Κοέλιο αναφέρθηκε στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, δεν θα πρέπει να κάνει κανείς ό,τι είναι δυνατόν να γίνει από τεχνικής άποψης και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση των δεδομένων. Διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ αρνητικό τρόπο τα δεδομένα αυτά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο συνάδελφος Άξελ Φως. Τα ε, δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρε ε, είναι προσωπικά δεδομένα. Μπορεί να είναι. Το αυτοκίνητό μου μαζεύει πολλά και διάφορα δεδομένα. Και όχι μόνο σχετικά με το αν ε, έχουν τελειώσει τα λάδια συλλέγει και δεδομένα σχετικά με το ε, ε, αν ε, τρέχω γρήγορα ή αργά, αν κάνω μεγάλες διαδρομές ή όχι, αν ξεκινάω προσεκτικά. Όλα αυτά τα δεδομένα συλλέγονται και το αργότερο όταν πάω στο γκαράζ μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι «Α, ορίστε μας, η ζύπλη πάντα τρέχει, πάντα ξεπερνάει το όριο της ταχύτητας». κάθε εξάμεινο ε, πρέπει να ε, αγοράζω καινούργια λάστιχα, αλλά πλημμυρίζει ε, το ταχυρομικό μου κουτί από προσφορές. Και μήπως τελικά η ασφαλιστική μου εταιρεία αυξήσει ε, τα ασφάλιστρα χωρίς να μου πει από πού έχει τα δεδομένα στο οποίο το στηρίζει αυτό. Μπορούν ε, λοιπόν ε, και τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρε να είναι προσωπικά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ψευδονιμοποίηση ή ανωνυμοποίησή τους. Θα πρέπει όμως και εδώ να είμαστε προσεκτικοί. Ε, και να αναφερθώ στο θέμα των ευφυών ε, ε, μετρητών, για παράδειγμα, για την κατανάλωση ρεύματος. Ο μετρητής μπορεί να διαπιστώσει ότι πιο πολύ ρεύμα χρησιμοποιώ Παρασκευή πρωί. Για ποιον, για ποιον σκοπό όμως να το γνωρίζει αυτό ο πάροχος ρεύματός μου. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πότε έχω τη μεγαλύτερη κατανάλωση, όχι όμως ε, αν ε, την χρησιμοποίησα για να κάνω ντους ή αν επειδή ε, έχω ανάψει τρεις τηλεοράσεις ταυτόχρονα. Διότι αν τα μόνα δεδομένα που συλλέγονται είναι ε, σε ποιο μέρο τη πόλη υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση, ποιε ώρε, τότε δεν χρειάζεται να ασχοληθώ εγώ με την ψευδονιμοποίηση ή την ανωνυμοποίηση. Και μια τελευταία παρατήρηση και συγγνώμη που μαγρικόρω. Ε, προκύπτουν εδώ και ηθικά θέματα. Υπάρχει θέμα όπως είναι η αυτόνομη οδήγηση. Αν λοιπόν εγώ δεν παρεμβαίνω καθόλου, Ε, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται πια να κάνω ε, την επιλογή από το αν ε, θα πατήσω την γιαγιά που περνάει το δρόμο ή αν θα σκοτωθώ μόνη μου επειδή θα την αποφύγω και θα τρακάρω σε ένα δέντρο ή αν η εναλλακτική λύση είναι να πατήσω ένα παιδάκι. Επειδή λοιπόν ε, με την αυτόνομη οδήγηση μόνο τον ε, οδηγό μπορεί να προστατεύσει κανείς, ε, αποτελεί αυτός προτεραιότητα και ποιος ξέρει ποιον θα πατήσει το αυτοκίνητο. Και τέλος, με την έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να παραπέμπουμε σε μια παλιά οδηγία για την προστασία των δεδομένων. σύντομα έρχεται το 2018, θα πρέπει λοιπόν να ε, παραπέμπουμε στο, ε, στη δέσμη των μέτρων ε, για την προστασία των δεδομένων. Thank you very much. Κύριε Μπόρη, σας ευχαριστούμε για αυτήν την έκθεση που προετοιμάσατε, Άννα, γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε σε ποιο πλαίσιο κινούμαστε εξετάζουμε το ζήτημα των μαζικών δεδομένων στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και βρισκόμαστε επίσης στη, χρονική στιγμή όπου ξεκινάει να εφαρμόζεται ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί η ίδια η διαδικασία αυτή της έναρξης εφαρμογής του κανονισμού ε, δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Επίσης, Τώρα ξεκινάμε ταυτόχρονα την αναθεώρηση της ε, οδηγίας e-privacy για την ιδιωτικότητα ε, στο ίντερνετ και τα ζητήματα της, εμπιστευτη... Ε, Τα ζητήματα λοιπόν τη ιδιωτικότητα και τη προσαρμογή στην τοποθεσία του χρήστη θα πρέπει να τεθούν γιατί είναι σχετικά και με το, αυτή την οδηγία και με την υπράγαση. Ε, έχουν επίσης τεθεί και άλλα ζητήματα για την ανοιχτή πρόσβαση στα ε, επιστημονικά δεδομένα, τη δημιουργία ενός ε, ε αποθετηρίου κεντρικού, ενός υπολογιστικού νεύσου, για το οποίο θα μπορούν οι επιστήμονες από την Ευρώπη να ανταλλάσσουν δεδομένα. Είχαμε συζητήσει και έχουμε ακούσει από εισηγητές από αυτή, την επιτροπή αλλά και σε άλλες επιτροπές ε, ζητήματα που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα η ρομποτική και αυτά πιστεύω πρέπει να αναφερθούν σε αυτήν την έκθεση. Βεβαίω πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα των πικτάτα από την πλευρά των θεμελιωδών δεδομένων βεβαίω χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που να ε, εμπνέει την εμπιστοσύνη, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι δεν είναι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Υπάρχει πολύ μεγάλος ποσοστό των δεδομένων που είναι διαθέσιμα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες που θα, ε, στους οποίους θα απόκειται η επεξεργασία τους θα είναι διαφορετικοί έτσι ώστε να μην περιορίσουμε την επιστημονική έρευνα. Ο Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ. Ε, πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση, να πω ότι το κείμενο της Άννα είναι μια πολύ καλή ε, βάση για να ξεκινήσουμε ε, τη συζήτησή μας για αυτό το ε, σημαντικό θέμα της σχέσης των Big Data με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τίθεται και ζητήματα διακρίσεων, τα οποία έχουν όντως τα πραγματεύεται το κείμενο ικανοποιητικά. Εγώ συμφωνώ πολύ με τον συνάδελφο ε, Μπόνι ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρη η διάκριση ανάμεσα στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μη προσωπικού χαρακτήρα, τα άλλα δεδομένα. Γιατί χρησιμοποιώντας ανωνυμοποιημένα, ανώνυμα δεδομένα θα μπορούσε, κανείς, θα μπορούσε να επιτρέψει κανείς πολύ μεγαλύτερη επεξεργασία. Ενώ στον τομέα των προσωπικών δεδομένων υπάρχει η αρχή της ελάχιστης χρήσης, που, της χρήσης του ελάχιστου ποσοστού των δεδομένων που είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας. Ε, ε, υπάρχει ήδη μια αντίφαση στο να μιλάει κανείς για τη χρήση των τεχνικών big data για την εφαρμογή και την εφαρμογή τους στα προσωπικά δεδομένα. Ε, ήδη από τις αρχές που έχουμε στο δίκαιο το ευρωπαϊκό δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια μαζική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, γιατί η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται πάντα ε, στο βαθμό που αυτή είναι απαραίτητη για την επίτευξη ενός νόμιμου σκοπού. Επομένως, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τις προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη νέων τεχνικών και καλύτερων τεχνικών ανωνυμοποίηση. Ε, ή ακόμα και την επιχειρηματική αξιοποίηση ε, της, αυτής της τεχνικής της ανανομοποίησης. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να κλείσει τη συζήτηση. Κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις τους. Και αναμένω να δω και τις τροπολογίες που θα προτείνουν. Πολλοί συνάδελφοι είπαν και συμφωνώ ότι θα χρειαστεί να συζητήσουμε με τους διάφερους ενδιαφερόμενους φορείς, δηλαδή εταιρείε ή φορείς που χρησιμοποιούν ήδη big ε, αλλά και άλλες και, και άλλους, όπως για παράδειγμα τις διοκτικές αρχές που είπε ο Μάριο, για να όπως η συνάδελφος Μαρία, για να συζητήσουμε μαζί του όχι μόνο τις, ευκαιρίε ε, που ε, έχουν εντοπίσει τη χρήση των Big αλλά επίσης και τα προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποδεχθούμε με κατεβασμένα τα χέρια και χωρίς να το σκεφτούμε ότι ζούμε σε μια οργολική κοινωνία και έτσι έχουν τα πράγματα και απλώς θα συλλέγονται όλα και περισσότερα δεδομένα που μας αφορούν. Ίσως να υπάρχει και μια δυνατότητα να δούμε αυτή την κατάσταση σαν μια ευκαιρία, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Ίσως να υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θα τα επιτυχαίναμε αλλιώς, παρά μόνο με τη χρήση των μαζικών δεδομένων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να, μπορούσε να αξιοποιηθεί η τεχνική του Big Data για να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις ή η δημόσια διοίκηση. Σκεφτείτε το σκάνδαλο των ε, Panama Papers, των εγγράφων του Παναμά, που είναι από τη φύση τους ε, μια μεγάλος, μεγάλος όγκος δεδομένων που ε, έτυχαν επεξεργασίας. Αναφέρθηκε και ο πρόεδρος σε αυτό μόλις τώρα. Θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα μπορούσε να ε, συνδεθεί η χρήση της ανωνυμοποίησης με συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, οικονομικής δραστηριότητας. Αλλά εγώ θέλω να είμαστε και ρεαλιστές. Κάνοντας, συσχετίζοντας κανείς διαφορετικές βάσεις δεδομένων ή σύνολα δεδομένων, είναι πολύ συχνά εφικτό να αξιοποιήσει κανείς πολλά ανωνυμοποιημένα δεδομένα και παρόλα αυτά να ταυτοποιήσει το πρόσωπο που τελικά ε, αφορούν τα στοιχεία αυτά. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονό ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Πρέπει να έχουμε αυτή τη γνώση για να τα καταφέρουμε να τα ρυθμίσουμε. Τις προάλλες είχα μια συνάντηση με εκπροσώπους ε, της των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και μου εξήγησαν πώς μοιράζονται τις, τα στοιχεία που έχουν εκείνη στη διάθεσή τους που αφορούν σε αυτοκίνητα με μια ασφαλιστική. Και μετά η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα και να αποφασίσει, για παράδειγμα, να μην δεχτεί να ασφαλίσει έναν συγκεκριμένο πολίτη αν βλέπει ότι έχει μια ιδιωτική συμπεριφορά που δεν τη κάνει. Επομένως, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους αυτούς και τις πρακτικές που ακολουθούνται και θα πρέπει να είμαστε αυστηροί και θαραλέοι με τον ίδιο τρόπο που κινηθήκαμε και ε, στην κατάρτιση του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων, του DPR. εκεί διαπιστώσαμε ότι οι επιχειρήσει του κλάδου καλωσόρισαν τον Γενικό Κανονισμό προστασία Δεδομένων γιατί ήταν η πρώτη φορά που γινόταν μια προσπάθεια να τεθεί ένα πλαίσιο κανόνων. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε και σε συνεργασία όλοι μαζί να έχουμε αυτή την θαραλέα και τολμηρή προσέγγιση ε, στο ζήτημα της ανωνυμοποίησης, ψευδονυμοποίησης και όλων των άλλων ε, εχεγγύων που μπορούμε να ε, επιβάλλουμε. Χαίρομαι επίση για την αναφορά που έκανε συνάδελφο στο ζήτημα τη εκπαίδευση. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τι διακυβεύεται, ποιοι είναι οι κίνδυνοι Ανέφερε επίση και την ε, συμμετοχή που θα πρέπει να έχουν οι, αρχές, οι εθνικέ αρχέ προστασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη-μέλη, ο συνάδελφος Κοελίου. Και κάτι ακόμα που ανέφερε ο συνάδελφος Μπόνι. είναι το ζήτημα της προέλευσης των δεδομένων και της, της βιογραφικής τοποθεσίας στην οποία ε, βρίσκονται οι βάσεις δεδομένων. Έχουμε μία τάση να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι με το τι κάνουν οι αμερικανικές εταιρείε με τις βάσεις δεδομένων τους. Αλλά για παράδειγμα για τις βάσεις δεδομένων που χτίζονται, που δημιουργούνται στην Κίνα, δεν έχουμε επιδείξει την ίδια, το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια ευαισθησία. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την πολύ σημαντική τεχνική υποστήριξη που μου, έδωσαν, καθώς επίσης και ε, τους συναδέλφους που βοήθησαν για να φτάσουμε σε αυτό το προσχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσω ότι η ακρόαση για το θέμα θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 15 Δεκεμβρίου, 3 ε, η ώρα. Περνάμε στο επόμενο σημείο τώρα στην ημερήσια διάταξη η Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται στην πρόληψη, ε, έρευνα, ε, εντοπισμό και δίωξη ποινικών ε, αδικημάτων. Πρόκειται για τη Συμφωνία Ομπρέλα το ε, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2016 το Κοινοβούλιο έλαβε έτοιμα σύμφωνης γνώμης από το Συμβούλιο βάσει των άρθρων 16 και 218 παράγραφος 6 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ω εισηγητής θα σας παρουσιάσω τώρα το σχέδιο σύστασης και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους και οι εισηγητές για τις παρατηρήσεις τους και φυσικά και σε όποιο άλλο μέλος ε, θέλει να παρέμβει. Λοιπόν, η συμφωνία αυτή ε, μας διαβιβάστηκε το Σεπτέμβριο, αλλά επίσης ε, υπάρχει και μια ιστορία πίσω από αυτήν. Το 2010, όταν ε, έγινε μια πολύ έντονη συζήτηση για το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του προγράμματος εντοπισμού των ΗΠΑ και την πιθανή συμφωνία μας για να νομιμοποιήσουμε τη μεταφορά στοιχείων στο σύστημα αυτά και τη συμφωνία για το αμερικανικό PNR, τα στοιχεία των επιβατών, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών προς συγκεκριμένα ζήτησε πάρα πολλές φορές μια συμφωνία ομπρέλα υπό τη σκέπη της οποίας θα υπάρχει επίπεδο προστασίας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ανθρώπων, προστασία δεδομένων και ιδιωτική ζωή όταν διαβάζονται δεδομένα ε, στον τομέα της έρευνας, της πρόληψης, ε, του εντοπισμού και της δίωξης ποινικών αδικημάτων στα πλαίσια της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά διζητήματα. Επομένως, ε, ε, δεν θα χρειάζεται στη συνέχεια να γίνεται διαπραγμάτευση για τα πρότυπα αυτά σε κάθε συμφωνία εκ του μηδενός, αλλά θα υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας, το οποίο θα ισχύει πάντα. και επομένως θα συμπληρώσει και τις ε, κείμενες συνθήκες ε, για τη, κυρίως ε, συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής και συμφωνίες που μόλις σας ανέφερα. Το Μάρτιο του 2011, στις 28 Μαρτίου πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις βάσει ε, μιας εντολής ε, που ενέκρινε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2010. Έκτοτε ε, γίνονταν διαπραγματεύσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, όπου μονογράφηκε η συμφωνία και τον Ιούλιο φέτος το Συμβούλιο αποφάσισε ε, επί της συμφωνίας ε, και την έστειλε για σύμφωνη γνώμη προς, την ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εισηγητής προτείνω βάσει και πολλών συζητήσεων και ανταλλαγών απόψεων που είχαμε με τους και οδησηγητές και με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και άλλες πλευρές, όπως για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας ε, για την συμφωνία αυτή. Θεωρώ ότι αποτελεί πολύ σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις ε, εγγυήσει για την προστασία των δεδομένων στα πλαίσια της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου μεταξύ των κρατών μαλλών και τις αρχές επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν ε, υπάρξει βέβαια και κάποιες ανοιχτές ερωτήσεις ε, στη διάρκεια της προηγούμενης ε, χρονιάς μετά τη μονογραφή της συμφωνίας, κυρίως από την νομική υπηρεσία για τρία ζητήματα. Το ένα αφορά το κατά πόσον η συμφωνία αυτή θα μπορούσε ίσως να ερμηνευτεί ως νομική βάση για μεταφορά στοιχείο ή ε, μπορεί να είναι απλώς ε, νομική βάση για να δίνει απόφαση καταλληλότητας, διότι η προστασία δεδομένων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της νομοθεσίας προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Μετά από τις ανταλλαγές απόψεων που έγιναν, είμαι πεπισμένος ότι δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως νομική βάση, αλλά χρειάζεται πάντα είτε ευρωπαϊκό δίκαιο είτε κάποια διεθνή συμφωνία για να ε, δοθεί έγκριση, έγκριση για κάποιες ε, μεταφορές δεδομένων. Επίσης, ε, είμαι ικανοποιημένος με τις εξηγήσει που μας δόθηκαν, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το ρόλο αυτής της συμφωνίας εν των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Πρέπει ε, να θεωρήσουμε ότι προστατεύει επαρκώς. Παρόλα αυτά, επέμεινα η διευκρίνηση αυτή να μην διατίθεται μόνο σε εμά, αλλά να δημοσιοποιηθεί μέσω επίσημης δήλωσης, η οποία ε, θα γίνει στα πλαίσια της έγκρισης αυτής της συμφωνία, ώστε ε, κάθε ε, μέρος ε, και φυσικά τα συμβολά με ένα μέρη της συμφωνία να γνωρίζουν σαφώς ότι αυτή είναι η ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ισχύει και για το δεύτερο σκέλος, δηλαδή το κατά πόσον η συμφωνία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και με κάποιες προσαρμογές ε, στο αμερικανικό δίκαιο για κάποιες εξαιρέσεις. Βάσει συγκεκριμένες πράξεις ε, που, πράξεων που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για τα δεδομένα PNR και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς που καλύπτει, που ε, καλύπτει επίσης και τη μεταφορά δεδομένων PNR και να είναι σαφές ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουμε ότι θα γίνουν αυτές οι κινήσεις και φυσικά ε, η συνέπεια είναι ότι εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, η συμφωνία αυτή δεν θα εφαρμόζεται πλήρως από την άλλη πλευρά και επομένως δεν θα ισχύει και σε άλλες διατάξεις από πλευράς μας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν αποτελεί κατάλληλη εγγύηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μπορούν πάντα να γίνονται έλεγχοι από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα πάντα είναι βάση της συμφωνίας και αν υπάρχουν οι εγγυήσει για την προστασία των δεδομένων, γεγονός που σημαίνει ότι οι εξισίες των αρχών προστασίας δεδομένων και ε, ε, κυρίως αυτών δεν περιορίζονται μέσω της συμφωνίας. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, μια διευκρίνηση, η συμφωνία αυτή καλύπτει και δικαστικές ε, διεκδικήσεις Δυνατότητες λοιπόν ε, για προσφυγή ε, στα δικαστήρια, κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και βάσει της πράξης για τη δικαστική προσφυγή που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2016 από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλύπτει δυνατότητες μόνο ε, για κάποιους φορείς ε, που ε, γίνονται σεβαστοί από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να μην καλύπτονται από την απόφαση λόγω συγκεκριμένων χωρών που καλύπτονται από το ε, πλευρά των ΗΠΑ. Εμείς θεωρούμε ότι τουλάχιστον για τους σκοπούς αυτής της συμφωνίας πρέπει να καλύπτονται όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι πολίτες τους κατά συνέπεια και ε, για τα άτομα τα οποία μόνιμα διαμένουν στις ε, χώρες μέλη και που δεν διαθέτουν ηθαγένεια. Εκεί υπάρχει ένα κενό και ελπίζουμε να επιληθεί και γι' αυτό ακριβώς και θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ε, κατά την εφαρμογή και τη συνέχεια αυτής της συμφωνίας θα πρέπει να εγκαταστεί σαφές ότι θέλουμε να καλύπτονται και αυτά τα άτομα στο μέλλον με πλήρη δικαιώματα και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Με αυτά λοιπόν νομίζω ότι και λόγω του γεγονότος ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν ε, βρίσκονται στην ίδια ακριβώς γραμμή πλεύσης ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλουν να καλύψουν όλους τους κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αυτή την περίπτωση δυνατότητας ε, προσφυγής. Η συμφωνία αυτή αποτελεί προστιθέμενη αξία και μια επιπλέον εγγύηση για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως θεωρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση εάν δεν καλύπτει τους πάντες θα μπορούσε να παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θεωρώ ότι τα πάντα καλύπτουν προκύπτονται από αυτέ τι ε, εξηγήσει, προτείνω λοιπόν να δοθεί η σύμφωνη γνώμη μα και από εκεί και πέρα να ε, θεωρήσουμε ότι αυτό αποτελεί και αφετηρία για άλλες ε, αντίστοιχες συμφωνίες και σε θέματα προστασίας δεδομένων και θεμελιωδών δικαιωμάτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να υπάρχει ένα κοινό πρότυπο και όχι διαφορετικά πρότυπα και αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων, διότι δεν θεωρώ ότι ε, επαρκούν πλέον για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Δύο μέλη έχουν ήδη ζητήσει το λόγο. Βλέπω βέβαια και κάποιους άλλους. Ο Άξελ Βος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι με όλη αυτή τη συζήτηση για την προστασία των δεδομένων, για τον κανονισμό, για την οδηγία, για τον ασφαλή λιμένα, για τη συμφωνία ομπρέλα, ε, έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε και κάποια πράγματα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και με βάση τη συζήτηση που είχαμε κάνει και τις διευκρινήσεις που είχαμε κάνει, νομίζω ότι έχουμε πετύχει πολλά. Όσον αφορά λοιπόν αυτήν την συμφωνία ομπρέλα, νομίζω ότι έχουμε πολλά άλλα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων μέχρι ε, να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στα πράγματα οι οποία να μπορεί να πρέπει να ενσωματωθούν. Τις ιδιαιτερότητες μπορούμε πάντα να τις προσθέσουμε εκ των υστέρων δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, αλλά έχουμε ένα καλό πλαίσιο και έχουμε καταβάλει νομίζω σημαντικές προσπάθειες και το περιγράψατε ακριβώς αυτήν την συμφωνία ομπρέλα μπορούμε να την εγκρίνουμε με ήσυχη τη συνείδησή μας. Έχουμε πετύχει πολλά και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και αυτό το βήμα. Το ΕΛΚ στηρίζει τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει το πλαίσιο αυτό να θεσπιστεί σύντομα. Και άλλωστε το μόνο εντό αγωγικών θέμα που ρυθμίζεται εδώ είναι η ανταλλαγή δεδομένων ε, μεταξύ ε, διαφόρων αρχών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή η συμφωνία αυτή την οποία μπορούμε να υπερψηφίσουμε με ήσυχη τη συνείδησή μας. Ευχαριστώ πολύ, Μαρή Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σημαντική στιγμή στις εργασίες μας, διότι ξέρουμε πόσο δύσκολη ήταν όλη η διαδικασία και όλη η συζήτηση. Στην ομάδα επίσης ε, και στην ομάδα εργασίας ε, συζητήθηκε το αποτέλεσμα αυτό. Και διαβάζοντας ε, το συμπέρασμα του εισηγητή, ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ανταλλαγή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι συμφωνούμε με αυτό. Έχουμε έτσι νέες εγγυήσεις ε, κατά την ε, ανταλλαγή δεδομένων. Ε, δεν είχαμε στο παρελθόν τέτοιες εγγυήσεις. Αυτό λοιπόν αποτελεί σημαντική πρόοδο. Επίσης, είχαμε αρκετά σημαντική συζήτηση σχετικά με τις ε, δικαστικές προσφυγές. Στην πράξη θα μπορούσε να έχουμε διάκριση ανάμεσα στους ε, υπηκόους και μη υπηκόους και αυξάνεται το ποσοστό υπηκών τρίτων χωρών, ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, στα κράτη-μέλη. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα κάποια στιγμή. Σημαντικό είναι να φροντίσουμε και η άλλη πλευρά ε, να μην ερμηνεύσει την ε, συμφωνία αυτή ως μέσο για να ε, επιτρέψει την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Μία χώρα θα μπορούσε δηλαδή να αρνηθεί να διαβάσει ε, τα δεδομένα επειδή πρόκειται για δεδομένα μη υπηκόων. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος κατάχρησης ε, και έλλειψης ε, δυνατοτήτων προσφυγής. Εάν λοιπόν φροντίσουμε οι αρχές προστασίας των δεδομένων να μπορούν να παρέμβουν, θα μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της συμφωνίας και να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ε, έχουμε τις ε, περιοδικές εκθέσεις και νομίζω ότι ήδη σε τρία χρόνια θα μπορέσουμε να κρίνουμε πώς θα λειτουργήσει η συμφωνία. Η γενική συζήτηση στην ομάδα μας μας έφερε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την συγκατάθεση, διότι όπως είπαμε δεν είναι η ιδανική λύση, είναι η καλύτερη όμως από όλες τις ε, ρεαλιστικές λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε για την σωστή εφαρμογή της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Σοφή Νετφέλτ από την Άλτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά θέλω να πω για τη συμφωνία αυτή. Καταρχάς έχουμε την ιστορία της. Κάποιοι από τους παρόντες θα θυμούνται ότι ήμουν μία από τους πρώτους ε, που ζήτησε ε, διατλαντική συμφωνία για την προστασία των δεδομένων. Είναι καλό λοιπόν που την έχουμε. Υπάρχουν επίσης νέα εχέγγυα και μάλιστα ε, διεύρυνση του δικαιώματος ε, για δικαστική προσφυγή. Όλα αυτό αποτελούν πρόοδο σίγουρα, αλλά ο διάβολος ε, υπάρχει στη λεπτομέρεια. Όσον αφορά λοιπόν τη διαδικασία, πρέπει να πω ότι καταρχάς με εκπλήσει που το χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση της έκθεσης αυτής. Ε, δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε γκρίνει έκθεση μέσα σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες. Σήμερα, 8 Νοεμβρίου, βλέπουμε την πρόταση ε, και 1η Δεκεμβρίου προβλέπεται ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ε, πριν από την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων ε, συζητούσαμε το θέμα αυτό επί 10 χρόνια. Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε επίγουσα διαδικασία αγνοώντας όλες τις νομοθετήσει που έχουμε λάβει από την νομική υπηρεσία, από την ομάδα εργασία ε, και από διάφορους άλλου άλλους φορείς. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. και γιατί όλοι διαμαρτύρονται για συμφωνίες όπως η ΣΥΤΑ, ε, ενώ εάν θεωρείτε την ΣΥΤΑ κακή, αυτή η συμφωνία είναι ακόμα χειρότερη. Ε, δεν καταλαβαίνω λοιπόν ούτε τα ε, διπλά μέτρα και σταθμά, ούτε τη βιασύνη. Όλοι λένε ότι δεν αποτελεί ε, ε νομική βάση για την διαβίβαση δεδομένων. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ε, νομίζω στο άρθρο 5.3 της ε, συμφωνίας, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, λέει ότι αν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, θεωρείται ότι ε, έτσι θεωρείται ότι έχουν επαρκή εχέγγυα, το οποίο σημαίνει κύριε εισηγητά στην πράξη ότι πρόκειται για μια ελευκό έγκριση. Και θα ήθελα να ακούσω την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι αν δεν πληρούνται εδώ τα κριτήρια σχετικά με τα απαραίτητα εχέγγυα, τότε τι επιπλέον εχέγγυα θα ζητηθούν πέρα από τη συμφωνία αυτή. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα. Στην πράξη λοιπόν έχουμε εδώ εν λευκό συμφωνή, ε, έγκριση για την ε, διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις Πολιτείες για τον σκοπό επιβολής του νόμου. Είμαι πολύ καιρό εδώ. Ε, οι, αναθεωρήσεις δεν αξίζουν ούτε το χαρτί πάνω στο οποίο έχουν γραφτεί. Ε, δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε ένα παράδειγμα που μία αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε για να ε, προσαρμοστεί να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας ε, θα ισχύει για όλη την αιωνιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι κάνουμε. Όσον αφορά λοιπόν την απόφαση περί επάρκειας, πρόκειται για εν λευκό επιταγή και ναι, μεν ε, υπάρχουν, ε, εδώ υπάρχει το θέμα της ε, δικαστικής προσφυγής, αλλά δεν ισχύει για τους μη υπηκόσους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην συνθήκη λέει ότι δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε διεθνείς συμφωνίες που να μην ευθυγραμμίζονται με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα και δεύτερον που είναι επίσης σημαντικό στο οποίο δεν δόθηκε πολύ προσοχή. Το δικαίωμα για δικαστική προσφυγή χορηγείται μόνο σε ανθρώπους σε συγκεκριμένες χώρες. Πώς Ισχύει αυτό λοιπόν για μια χώρα εφόσον ε, συμφωνεί στην ανταλλαγή δεδομένων για, προσέξτε με, εμπορικούς λόγους. Έχουμε λοιπόν μόνο το θεμελιώ δικαίωμα ε, δικαστικής προσφυγής αν είμαστε διατεθειμένοι να ε, διαθέσουμε τα δεδομένα μας στην Google για εμπορικούς σκοπούς. Πραγματικά εγώ δεν βλέπω να συνάδει αυτό με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και πείτε μου ότι είμαι κοινική. πείτε μου ότι δεν έχω εμπιστοσύνη, αλλά η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχουμε εδώ παρόν τον κύριο ε, Σιγαρέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχτηκε ότι όλο αυτό το θέμα βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα ε, ανακαλέσουν, θα αποσύρουν ε, τις παρεκκλήσεις που ισχύουν για κάποια προγράμματα οι πιθανότητε όμω να συμβεί αυτό είναι μηδενικέ. Αυτό θα συμβεί όταν δείτε γρούνια να πετάνε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ποτέ δεν θα ε, ε, ανακαλέσει αυτέ ε, τι παρεκκλήσει. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου επιβεβαιώσει αυτά που άκουσα. Σε μια ανεπίσημη συνάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ότι ναι, το ξέρουμε, αλλά Η συμφωνία αυτή δεν ε, θα ε, ισχύει νομικά, αλλά εμείς ε, θα προχωρήσουμε και αν δεν αρέσει στους πολίτες να πάνε στα δικαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν αυτό είναι αλήθεια, είναι διατεθειμένη εσκεμένα να συνάψει συμφωνία που δεν έχει νομική ισχύ και αφήνει τους πολίτες να προσφύγουν στα δικαστήρια. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται ε, το κράτος δικαίου, ε, τις συνθήκες ε, και το δικαστήριο, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ πέρα. Λέτε ότι θέλετε να τα λύσετε όλα προσθέτοντας μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λύση στη συμφωνία ΣΥΤΑ ενώ μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εδώ. Αλλά πέρα από αυτό μια τέτοια δήλωση δεν λύνει τίποτα. Εάν η συμφωνία αυτή καθ' αυτή ε, δεν είναι στεγανή, δεν θα μπορέσουμε ε, να την λύσουμε με προσκοπικό όρκο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν ε, με μια απλή διακήρυξη. Οι εξαιρέσει από τον νόμο περί ιδιωτική ζωής θα πρέπει να ανακληθούν. Θα πρέπει η συμφωνία αυτή να συνάδει με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και εγώ είμαι πεπισμένη, αλλά ευχαρίστω θα ακούσω συμβουλές από οποιονδήποτε γνωρίζετε καλύτερα τα θέματα αυτά από μένα, εγώ πάντως ε, δεν βλέπω πώς μπορούμε να συνάψουμε συμφωνία που δίνει δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε αντάλλαγμα υπόσχεσης από τα κράτη-μέλη ότι θα δίνουν δεδομένα στι Ηνωμένε για εμπορικούς σκοπούς. Και κύριε Ισηγητά, μία ακόμα παρατήρηση, διότι υπάρχει άλλη μια προϋπόθεση για την δικαστική προσφυγή. Συγγνώμη, ε, αναδιατυπώνω. Η διαβίβαση δεδομένων στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ε, στην, ε, στο Privacy Shield που υιοθετήθηκε πρόσφατα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα νομικά μέσα, αλλά αυτό είναι το κυριότερο από αυτά. Εσείς, όπως και εγώ, είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά αυτό το Privacy Shield. Εάν λοιπόν Ε, ακυρωθεί, αν προσφύγει κάποιος στο δικαστήριο, τότε θα καταρρεύσει άλλος ένας πυλώνας αυτής της συμφωνίας. Η υπόσχεση αυτή, λοιπόν, μάλλον η απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διαβιβάσουμε δεδομένα για εμπορικού σκοπού ε, μπορεί μόνο ε, να τηρηθεί με, τι να σας πω, με άλλους τρόπους. Ε, τι να σας πω, όλο αυτό εδώ πέρα είναι ένα τρομερό μπέρδεμα, η ομάδα μου δεν είναι διατεθειμένη να τη στηρίξει και θα πρέπει οι τροποποιήσεις να είναι τέτοιες ώστε να έχουμε ένα στενανό κείμενο, πάντως όσα έχει αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Thank you very much. Uh, the next is Ernst for Group. Σας ευχαριστώ για την ομάδα ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό, ε, καλός ή κακός, ε, και τώρα το θέμα είναι αν θα δηλώσουμε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Τι να σας πω, δυστυχία νιώθω και δεν μπορώ να σας πω ότι με ήσυχη τη συνείδηση και χωρίς αφέλεια μπορώ να συμφωνήσω με αυτά ε, που υπάρχουν εδώ στο έγγραφο. Όλα είναι υπέροχα. Η συγητή λέει ότι σημαντικό είναι να πούμε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν αποτελεί την νομική βάση για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Ναι, ωραία, αυτό το βρίσκω αξιέπαινο, αλλά το θέμα είναι πώς θα το δει αυτό η άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε με όλη την αιτιολόγηση. Συμφωνώ με όλη την αιτιολόγηση, αλλά ε, δεν έχω κάποια εγγύηση ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, πράγματι θα ενεργήσουν σύμφωνα με αυτά που λέγει εδώ. Επίσης, ε, η απόφαση περί επάρκειας, και αυτό συζητήθηκε επί μακρόν. Δεν έχουμε όμως εδώ πέρα σαφήνια και διαβάζοντας το κείμενο, ε, διαπιστώνω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε το σημείο αυτό. Και ε, όσον αφορά την περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων ε, και ε, τα, τις περιόδους διατήρησης. δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που έχουμε εδώ μπροστά μας. Ε, βρίσκω ότι είναι προβληματική η ρύθμιση. Δικαστική προσφύγη και αυτή είναι μια μακρά συζήτηση. Με λίγη τύχη να ισχύει για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για τους άλλους, μα μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να ισχύουν για όλους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε πράγματι με ήσυχη τη συνείδηση να υπερψηφίσουμε μια τέτοια συμφωνία και όπως πιστεύουμε στο Θεό, να πιστεύουμε ότι όλα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στην αιτιολόγηση θα οδηγήσουν σε καλό αποτέλεσμα. Ειλικρινά δεν μπορώ να δω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, θα πρέπει ε, στο διατακτικό του κειμένου να συμπεριλάβουμε ε, αυτά που ε, συμπεριλαμβάνονται στην αιτιολόγηση και να αποτελήσουν προϋποθέσεις. Αλλά ως έχει αυτή τη στιγμή το κείμενο, πιστεύουμε ότι οδηγεί σε μεγάλη ανασφάλεια και φοβάμαι ότι πρέπει να πούμε ότι ότι τι να κάνουμε αυτή τη συμφωνία έχουμε, δεν μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα παραπάνω, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Okay, thank you. Uh, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες Αγγελιά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αλλά πολύ σημαντικό. Έχουν ήδη υποθεί πολλά. Και εγώ θα συμφωνήσω με τη δικιά σας ε, ανάλυση που ήταν πολύ ενδελεχής με την ιδιότητα συγητής. Αλλά επίσης θα συμφωνήσω και με τους συναδέλφους που έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για ορισμένα θέματα. Και άρα, εγώ θα ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια ρήτρα για την περιοδική αναθεώρηση της ε, και αξιολόγηση μάλλον της εφαρμογής της ε, συμφωνίας. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη σύμφωνη γνώμη του και η συμφωνία προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί το Δεκέμβριο, θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγεται ότι θα γίνεται αυτή αξιολόγηση περιοδικά, αναμένουμε αλλαγή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιανουάριο. Θα ήθελα να μου πείτε τι προβλέπετε για το κατά πόσον αυτή η αλλαγή της Αμερικανικής, ε, του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να έχει κάποια επίπτωση στην πιθανότητα να άλλαξει η Αμερικανική νομοθεσία και συγκεκριμένα το σημείο που αφορά στην δικαστική αξιολόγηση για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων που αφορούν Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό που υπονοώ είναι ότι αυτή η αλλαγή του Πρόεδρου των ΗΠΑ, εν πάση περιπτώσει, δεν θα οδηγήσει στο χειρότερο σενάριο, γιατί τότε με το χειρότερο σενάριο ε, σίγουρα θα υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες σε αυτά που σχεδιάζουμε. Και μάλλον απίθανο θα είναι, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν σοβαρά την συμφωνία. Αν όμως η εκλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι η... δεν οδηγήσει στη χειρότερη επιλογή, αλλά στην άλλη. Τότε Ποιος πιστεύει, το πιστεύετε ότι στην περιοδική αξιολόγηση και στο ρόλο επίσης που θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την αξιολόγηση. Γιατί εμείς δεν, χρειάζεται να έχουμε λόγο μόνο τώρα που, δίνουμε τη που θα πιθανώς να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας, αλλά και στο μέλλον, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή της περιοδικής αξιολόγησης της συμφωνίας. Επομένως, πολλά θέματα δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί όσον αφορά την διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να προωθήσουν αυτά που τους ζητούμε για την υιοθέτηση της συμφωνίας και για να καταλάβουμε τελικά τι σκοπεύει να κάνει με την περιοδική αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκπληρώσει το ρόλο του της και να, είναι, να λογοδοτεί εναντί του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα δώσω το λόγο τώρα στην εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στα ερωτήματα των συναδέλφων, τον κύριο Τζενκαρέλη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά να ευχαριστήσω εσάς, τον εισηγητή και τους κοιόδους εισηγητές και εν γέννη την Επιτροπή σας για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Το συζητούμε εδώ και χρόνια το θέμα αυτό. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά στο θέμα αυτό, τη βοήθειά σας, την προσπάθειά σας και τη συνεχή σας υποστήριξη που ήταν θεμελιώδη σημασία για να έχουμε συμφωνία ε, για το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δικαστική προσφυγή και δεν θα πρέπει να το θεωρείτε ως κάτι ίσονος σημασίας. Ε, δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που έχουμε συζητήσει, που έχετε ακούσει και από μένα. Ακούστηκε και το όνομά μου για αυτά που έχετε ακούσει από μένα στις διάφορες ανταλλαγές που έχουμε κάνει. Αλλά θα πρέπει να αναφερθώ στο εξής. Αυτή είναι η πρώτη φορά που όχι μόνο σε διατλατικό επίπεδο, αλλά γενικά σε διεθνές επίπεδο, έχουμε πλέον μια γενική συμφωνία προστασίας δεδομένων στο συγκεκριμένο τομέα της ε, ε, επιβολής του νόμου. Πρόκειται για κάτι λοιπόν το οποίο προσθέτει προστασία και δικλείδες ασφαλείας και αυτό είναι ε, άνευ προηγουμένου. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα φέρει άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές σε όλους τους υποκείμενους στα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η πλειοψηφία των διατάξεων αφορούν τους πάντες ε, και ε, υπηκόους και μη υπηκόους και ε, θα επανέλθω στο σημείο αυτό. άμεσα ωφέλη όσον αφορά τα δικαιώματα και την προστασία ε, για όλους τους υπηκόους και κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται ανταλλαγές ε, δεδομένων βάσει ε, υφιστάμενων συμφωνιών, ε, βάσει νόμων και μία από αυτές τις προστασίες δεν ισχύει. Έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προστασίες. Με αυτή τη συμφωνία τρόπον την αναφέρθηκε και αυτό, θα διορθώσουμε και τις ε, παρούσες ασυμμετρίες και λήψεις ισορροπίας που υπάρχουν ε, σε θέματα ε, προστασίας στον τομέα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων και από τις δύο πλευρές του Αυτή τη στιγμή οι πίκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών απολασβάνουν αυτή την ε, προστασία, αλλά τα δεδομένα των Ευρωπαίων μπορούν ε, να ε, μεταφέρονται για λόγους επιβολής χωρίς να απολαμβάνουν της ίδιες προστασίας. Επομένως, για να αναφερθώ και στο ψήφισμα του ίδιου του Κοινοβουλίου, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι τα δικαιώματα των Ευρωπαίων να μπουν επίσης επί με τα δικαιώματα των Αμερικανών και φυσικά δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Η συμφωνία θα πρέπει να προσφέρει και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου ε, στην συνεργασία επιβολής του νόμου. Για να γίνει αυτό, όσο πιο σύντομα τεθεί σε ε, ισχύ η συμφωνία ομπρέλα, τόσο πιο εύκολο θα είναι για μας ε, τους Ευρωπαίους τα πράγματα, τόσο πιο καλά μάλλον θα είναι. Ε, και αντιλαμβάνομαι φυσικά και αυτά το οποίο ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπενθύμησε και ο Πρόεδρος ε, και η συγητής σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό ακριβώς και Προσπαθούμε να έχουμε μία δήλωση η οποία θα ε, απαντήσει στα θέματα αυτά και θα δώσει και τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Πιο συγκεκριμένα, και αυτό άλλωστε μου δίνει και τη δυνατότητα να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια, ε, αν όχι και όλα, ε, για την φύση αυτής της συμφωνίας. Το πρώτο σημείο λοιπόν για το οποίο θα δώσουμε διευκρινήσεις είναι η φύση αυτής της συμφωνίας. Αυτό καθορίζεται από το κείμενο της συμφωνίας, δεν αποτελεί βάση για ε, μεταφορές είναι, δεν είναι μια συμφωνία η οποία προβλέπει γενικότερη έγκριση για μεταφορά δεδομένων. Το πεδίο εφαρμογής ε, της διάταξης για την ε, δικαστική προσφυγή. Και πάλι εδώ, σαφώς από το κείμενο προκύπτει ότι το άρθρο για τη δικαστική προσφυγή θα ισχύει πλήρως για τη μεταφορά δεδομένων PNR που βασίζεται στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών για τα δεδομένα των επιβατών. Όσον αφορά τη δυνατότητα άλλων μέτρων μέσων δικαστικής προσφυγής, αφορά όλους τους ε, κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ισχύουν, η δικαστική προσφυγή ισχύει μόνο για τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν άλλα μέτρα, ε, δυνατότητε προσφυγή που ε, καλύπτουν ε, όλους τους κατοίκου, ανεξάρτητα αν είναι υπήκοοι ή απλώ κάτοικοι τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, να μπορούν να ζητήσουν τήρηση των δικαιωμάτων τους και να λάβουν και τι απαραίτητε αποζημιώσει ή τα κατάλληλα μέτρα. Κάτι ακόμα το οποίο θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε είναι η εξουσία των δικών μας αρχών προστασίας δεδομένων ε, θα μπορούν πλήρες να ασκήσουν τον εποπτικό τους ρόλο, να ερευνήσουν, παρεμπιπτόντως ε, να πω ότι αναφέρονται ρητός ε, σε αρκετές διατάξεις της συμφωνίας αυτής. Θα υπάρχει ουσιαστικό στοιχείο και έχει ήδη συμφωνηθεί αυτό της συμφωνίας και υπάρχει η δυνατότητα να ερευνούν, να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν μεμονωμένες καταγγελίες. Ένα τμήμα της συμφωνίας και τμήμα της εφαρμογής της συμφωνίας είναι τι ε, προβλέπεται από πλευράς εποπτείας και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πιστεύουμε ότι αυτές οι διευκρινήσεις ε, διασκεδάζουν τις αμφιβολίες σας και ελπίζουμε να ε, ανοίξουν και δρόμο για θετική ψήφο από πλευράς Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ υπήρχε και μια παρατήρηση ακόμα που θέλει να κάνει Σόφη Ίνεμπελ, σύντομα όμως. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προώθηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν απαντήσετε στην ερώτησή μου. Σα δίνω ένα παράδειγμα και ε, σα παραθέτω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μου στείλετε εσεί. Αφορά την ανάγκη οι Ηνωμένε Πολιτείε να άρουν την εξαίρεση για το PNR και για όλα τα υπόλοιπα. Εσεί λέτε και σα παραθέτω. Με άλλα λόγια, προκειμένου να συμμορφωθούμε με αυτή τη συμφωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να τροποποιήσουν κάποιους εκτελεστικούς κανόνες και διοικητικέ πρακτικές. Εσείς τα λέτε αυτά. Εσείς μας λέτε ότι είναι απαλήτως απαραίτητο να γίνει αυτό. Και τώρα δεν απαντάτε. Όσον αφορά την ανταλλαγή εμπορικών δεδομένων. Στην πράξη για τη δικαστική προσφυγή λέει, δεν ξέρω και σε ποιο άρθρο είναι, όταν περιγράφει τι πρέπει να κάνει μια χώρα προκειμένου να θεωρείται ε, ε, αρμόδια χώρα. Καταρχά, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προστασία ιδιωτική ζωή για την ανταλλαγή δεδομένων με τι ΗΠΑ. Εντάξει. Δεύτερον, θα πρέπει να επιτρέπει τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων για εμπορικού σκοπού μεταξύ τη χώρα τη και των ΗΠΑ. Αυτή είναι από την ε, πράξη για την δικαστική προσφυγή. Δεν το έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου δεν είναι από κύμα της φαντασίας μου, επομένως θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Διότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται εδώ και μας παίζει την κασέτα συνέχεια για τα πράγματα που είναι καλύτερα από αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν η συμφωνία αυτή κατά 99% είναι εξαιρετική, υπάρχει ένα 1% που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, πολιτών που δεν είναι υπηκοί ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά διαμαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι καταπληκτικά. Τα πάντα είναι καλά, αλλά υπάρχει και το εξή. Σαν να παίρνουμε αυτοκίνητο και να μου λέτε τέλειο αυτοκίνητο, αλλά ένα λατωματάκι έχει, δεν έχει φρένα. Θέλω πραγματικά να μου απαντήσετε στην ερώτηση. Δεν θέλω να μου πείτε ότι προ το παρόν τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται για τα θεμελιώδη δικαιώματα και απλώ στέλνουν δεδομένα χωρί να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι στο επιχείρημα για να προσπαθήσετε να με πείστε για κάτι το οποίο δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Για να συνεχίσω και τη μεταφορά με το αυτοκίνητο, δεν λειτουργεί το αυτοκίνητο. Τρία χρόνια ρωτάω το ίδιο πράγμα. Ε, έχω κουραστεί. Συνέχεια και συνέχεια τα ίδια πράγματα σας ρωτάω. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει την ερώτηση, παρακαλώ. Πολύ χαίρομαι που η αλληλογραφία μας ε, ε, αποτελεί αντικείμενο συζήτηση, εν μέρη βεβαίω, γιατί αυτό που σας εξήγησα σε αυτό το μήνυμα και θα εξηγήσω και εδώ, είναι ότι υπάρχει μία διαφορά, υπάρχει μία σύγχυση. Καταρχάς υπάρχει σύγχυση μεταξύ του περιεχομένου της συμφωνίας και της σωστής εφαρμογής. Και βεβαίως για κάθε διεθνή συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή εφαρμογή. Τι έχει σημασία όμως όταν εξετάζουμε μια συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η συμφωνία αυτή δημιουργεί διεθνείς υποχρεώσεις. Θα είναι δεσμευτική για την άλλη πλευρά. Και σε αυτό το σημείο το κατά πόσον τα δεδομένα PNR θα καλύπτονται από την ε, δυνατότητα δικαστικής προσφυγής ε, βάσει της ε, διάταξης που υπάρχει. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο εργαλείο στο οποίο σας παρέπαμψα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο με συγκεκριμένη διάταξη σε αυτή τη συμφωνία και εάν, όπως και για άλλες διατάξεις αυτής της συμφωνίας, η σωστή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σημαίνει ότι η άλλη πλευρά θα πρέπει να τροποποιήσει κάποιες από τους κανόνες ή τις πρακτικές της, οι Ηνωμένε Πολιτείε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι και συνέπεια αυτή τη διεθνού υποχρέωση. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία για τη συζήτηση σήμερα είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη διεθνής υποχρέωση όλες οι μεταφορές δεδομένων που καλύπτονται από, αυτές τη, από αυτή τη συμφωνία να ε, καλύπτονται και από τα δικαιώματα δικαστικής προσφυγής. Η κυρία Ινετφέλτ, μία ερώτηση. Καλά και άγια όλα αυτά διότι βεβαιώνεται το ίδιο. Υπάρχει υποχρέωση από πλευρά ΗΠΑ και αν υπογράψουμε και εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία, υπάρχει υποχρέωση από πλευρά ΗΠΑ να άρουν την εξαίρεση για το PNR και αντίστοιχα προγράμματα. Και λέτε ότι αυτή είναι υποχρέωση και είναι τμήμα τη εφαρμογή. Όμω, από την εμπειρία που έχω εγώ μέχρι τούδε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν εποπτεύει τη σωστή εφαρμογή και ε, εξετάζει τις συμφωνίες, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι από τη στιγμή που θα αποφασιστεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πει «Α, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ήραν την εξαίρεση, δεν θα αναστείλουμε τη συμφωνία». Δεν θα το κάνετε. Στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτή η συμφωνία θα υπογραφεί, θα την αναθεωρήσουμε χίλιες φορές, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα άρουν την εξαίρεση και εμείς θα συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε αυτά. Αυτό θα γίνει και δεν θα γίνει με το όνομά μου. Okay. That's the commission wants to have δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει κάτι άλλο ή καλυφθήκατε. Να προσθέσω στην ε, προηγούμενη απάντησή μου ότι το θέμα της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας και πιο συγκεκριμένα της διάταξη που αφορά τη δικαστική προσφυγή είναι τόσο σημαντικό που η ίδια η συμφωνία λέει ότι η εφαρμογή της δικαστικής προσφυγής είναι ένα από τα ουσιαστικά ζητήματα της ετήσιας αναθεώρησης, της κοινή συγγνώμη άρθρο ως περαιτέρω επιβεβαίωση λοιπόν, και αυτό δεν είναι δήλωση, αυτό είναι αυτό ε, που έχουν ήδη συμφωνήσει οι διάφορε πλευρέ. Ούτε mail δικό μου, ούτε δήλωση δικιά μου. Επομένω, είναι ένα τομέα στον οποίο θα προσέξουμε ιδιαίτερα για την κοινή αναθεώρηση και σα καλώ επίση να διαβάσετε και το άρθρο για την αναστολή, το οποίο αναφέρεται στην παραβίαση Τη συμφωνία και τις συνέπειες τη παραβίαση αυτή τη συμφωνίας. Παρεπιπτόντω, πρόκειται για μία ακόμα πτυχή η οποία ε, θα ε, αντιμετωπίσουμε και στη δήλωσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω και πάλι το λόγο στον υποφαινόμενο ω εισηγητή και να απαντήσω και σε κάποιες από τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσει που, παρατηρήσεις που έγιναν. Η συμφωνία, όπως διαπραγματεύτηκε βεβαίως Βι- έτυχε διαπραγμάτευση ε, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, από το 8 ε, Δεκεμβρίου του 2015 και τα έχουμε στα χέρια μας πάνω από ένα χρόνο. Δεν πρόκειται ούτε για ταχεία διαδικασία, ούτε τίποτα άλλο. Έγιναν πολλές ανταλλαγές απόψεων, όπως γνωρίζετε, μεταξύ σχεδόν συγητών για το περιεχόμενο της συμφωνίας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έκθεση είναι πολύ απλή. Πρόκειται απλώς για τη σύμφωνη γνώμη μας. Ναι ή όχι θα πούμε, δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο και όπως επίσης γνωρίζετε, σε τέτοιες εκθέσεις είναι λογικό να γίνονται αυτά κατά αυτόν τον τρόπο. Ως προς την ουσία, η συμφωνία αυτή νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφής ε, ως προς την ουσία της και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Δεν αποτελεί νομική βάση για την ανταλλαγή, πουθενά δεν λέει ότι είναι νομική βάση, είναι απόλυτα σαφές και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου δεν το αμφισβητεί σε καμία περίπτωση αυτή δεν αποτελεί νομική βάση για τις, νομικές, ε, για τις ε, μεταφορές. Πρέπει πάντα να υπάρχει εθνικό δίκαιο, ενωσιακό δίκαιο ή εθνική ή ενωσιακή συμφωνία με τρίτη χώρα σε αυτή την περίπτωση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, το οποίο θα επιτρέπει να ε, γίνεται η μεταφορά. Αυτό που κάνει η συμφωνία είναι απλώς να δημιουργεί πρότυπα. Και αυτό παρεμπιπτόντως είναι και τεράστια διαφορά σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες. Στι εμπορικέ συμφωνίε γίνεται αμοιβαία αναγνώριση προτύπων, ε, αποδεχόμενο ότι μπορεί να έχουμε χαμηλότερε προδιαγραφέ στις αγορές Η συμφωνία αυτή δημιουργεί παρεπιπτόντως υψηλά πρότυπα και για τι δύο πλευρέ. Δημιουργεί κοινά πρότυπα, είναι τεράστια διαφορά και πολύ θα ευχαριστημένου θα ήμουν αν είχαμε τέτοιε συμφωνίε και στον τομέα του εμπορίου, αντί να έχουμε αμοιβαία αναγνώριση. Νομίζω ότι είναι τεράστια διαφορά και πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά την έγκριση, όπως σας είπα, σε καμία περίπτωση δεν δίνει έγκριση για οποιαδήποτε μεταφορά αυτή η συμφωνία. Επομένως, δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτή είναι έγκριση για οποιαδήποτε μεταφορά ε, ή ε, μία έγκριση γενικότερη. Σε καμία περίπτωση δίνει έγκριση για ε, μεταφορές, για παράδειγμα, η συμφωνία PNR ε, ή η συμφωνία TFTP. Αυτές είναι συμφωνίες αμοιβαίας ε, και νομικής συνδρομής. Οι περισσότερες από αυτές τις συμφωνίες έχουν πολύ χαμηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων και αυτή η συμφωνία θα συμπληρώσει αυτές τις παλιότερες συμφωνίες. Επομένως, έτσι θα φτιάξουμε τις παλιές συμφωνίες, οι οποίες παρεμπιπτόντως εφαρμόζονται τώρα και έχουν ψηφιστεί από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων εδώ στο Κοινοβούλιο. Αν ζητήσουμε να μην παραταθεί η δικαστική προσφυγή σε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε, εάν είναι απέτηση που κάνει παράνομη αυτή τη συμφωνία. Όλες οι συμφωνίες λοιπόν μεταφοράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι παράνομες διότι δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής προσφυγής σε καμία περίπτωση στις συμφωνίες αυτές. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι οι συμφωνίες αυτές είναι παράνομες λόγω αυτού. Κυρίως θα έλεγα ότι οι συμφωνίες μεταφορές για το PNR και το TFTP παραβιάζουν τη συνθήκη διότι δεν είναι αναλογικές. Αυτό είναι το, το ουσιαστικό. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό εδώ τώρα. Δεν υπάρχει έγκριση για καμία μεταφορά εδώ. Αυτό ε, απλώς αποτελεί κατάλληλη δικλίδα ασφαλείας και μια κατάλληλη δικλίδα ασφαλείας που, θεωρούμε, που θεωρώ ότι είναι δέουσα σε αυτή την περίπτωση. Προστατεύεται το νοσιακό δίκαιο σε αυτή τη συμφωνία. Φυσικά δεν θα έχουμε απόλυτα τον ίδιο τρόπο ρύθμισης με τρίτη χώρα, αλλά έχουμε τις υψηλέ προδιαγραφές που ζητά και το δικαστήριο και είναι και βάση τη συνθήκης, επομένως θα βελτιώσει όλε τι υπάρχουσες συμφωνίες και νομικέ βάσεις για μεταφορές δεδομένων και θεωρώ ότι αποτελεί άλμα με τις διευκρινήσεις, τις οποίες βεβαίως ακόμα ζητώ να ε, προσαρτηθούν σε αυτή τη συμφωνία όταν θα ε, δημοσιοποιηθεί στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και να ε, δηλωθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά ότι είναι απόλυτα σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική ερμηνεία. Και επίσης να πω ότι ακόμα κι αν υπάρξει κάποιο ερωτηματικό για το κατά πόσον οι Ηνωμένε Πολιτείε εφαρμόζουν πλήρως ε, τη συμφωνία, είναι απόλυτα σαφές ότι αν δεν την εφαρμόσουν, για παράδειγμα, στον τομέα των εξαιρέσεων για την ε, ε, πράξη για την ιδιωτική ζωή ή αν δεν προσφέρουν δικαστική προσφυγή σε ένα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για οποιοδήποτε λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε παραβιάζουν τη συμφωνία και τότε αυτό σημαίνει ότι από εκείνη τη στιγμή και πέρα δεν αποτελεί κατάλληλη εγγύηση. Επομένω, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε εγγύησει για κάθε μεταφορά από εδώ και πέρα και από όλα τα κράτη-μέλη. Με αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι πλήρως αιτιολογημένο να ε, προτείνουμε αυτή την άγουσα και θα είναι τεράστιο άλμα εάν καταφέρουμε να ε, δεχτούμε αυτή τη συμφωνία και στο μέλλον θα πρέπει να ζητάμε πολύ περισσότερες τέτοιες συμφωνίες και πρότυπα. Να ευχαριστήσω και όλους τους κοιόδης που συνεργάστηκαν μαζί μας για το θέμα αυτό τόσα χρόνια και βεβαίω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το διαπραγματεύτηκε αυτό εκ μέρου μας. Και ολοκληρώσαμε εδώ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 11 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Να ολοκληρώσουμε με το σημείο αυτό, γιατί έχουμε λίγα λεπτά. Ελπίζουμε να μας παραχωρήσουν διερμηνείς κάποια επιπλέον λεπτά, γιατί έχουμε άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση τη έκθεση τη Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την αποστολή τη Ηνωμένε Πολιτείε 16 με 20 Μαου 2016. Έξι συνάδελφοι από τη ΛΥΜΠΕ και εγώ ω επικεφαλής της αποστολές, ο Κλωτ Μωράε, και άλλοι συνάδελφοι ταξιδέψαμε στη Washington, στο Σαν Φρανσίσκο και στη Silicon Valley. Σε συνέχεια προηγούμενων αποστελών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ προς ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στόχος ήταν να έχουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες για το πώς έχει κατάσταση και πώς ε, προοδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής πολιτικών ελευθεριών, όπως ε, η ε, Συμφωνία για την Προστασία Δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή, η Συμφωνία Ομπρέλα, ε, εφαρμογή της νομοθεσίας, αντιποτόπιση της τρομοκρατίας, ριζοσπαστικοποίηση, στρατηγική, μέτρα τα οποία λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματα άρσης της απαλλαγής της υποχρέωσης θεώρησης. Πήγαμε στο Σαν Φρανσίσκο και στη Σινικόν Βάλεϊ και στη Ουάσιγκτον για να συναντήσουμε ενδιαφερομένους και ακούσαμε τις απόψεις τους για θέματα υψηλής σημασίας. Θα δείτε ότι ε, πρόκειται για πολύ ε, πυκνό πρόγραμμα με αρκετές συναντήσεις, γερουσιαστές, ενδιαφερομένους, ε, πανεπιστήμια το Πανεπιστήμιο του Στάντφορ, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο κλπ. Η Επιτροπή Λίμπε συζήτησε διάφορα θέματα και μπορέσαμε να έχουμε ενίσχυση τη συνεργασία με τις διοικητικέ αρχές των ΗΠΑ, με το Κογκρέσον και μια ειλικρινή ε, ανταλλαγή απόψεων. Να δώσω τώρα τα το λόγο στα μέλη τη αποστολή, εάν θέλουν να προσθέσουν κάτι. Roberta Thank you very much, um, um, uh, chair. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ευχαριστήσω και εγώ τη γραμματεία. Καθώς και το γραφείο μας στην Ουάσιγκτον που εκπώνησε τόσο εξαιρετικό πρόγραμμα. Πρώτη φορά μου ήταν στη Σιλικονβάλη και με ε, εντυπωσίασε το επίπεδο συζήτηση που είχαμε με τους ε, περί προστασίας δεδομένων ε, της Google και της ε, ε, Facebook. Θα ήθελα πολύ να είχαμε περισσότερες συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου Μέχρι τώρα ε, σε όλες τις ε, ε, επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχω διαπιστώσει ότι θα ήταν καλύτερο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο ποιοι θα είναι οι συνομιλητές μας να έχουν να κάνουν τα δικά μας θέματα όπως είναι η προστασία του ιδιωτικού βίου κλπ. πάντως. γενικά ήταν πολύ καλά οργανωμένη η αποστολή και προσλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε με τη νέα κυβέρνηση. Μία συζήτηση που θα πρέπει να ε, όπου θα πρέπει να σταθούμε λίγο είναι η συζήτηση που είχαμε με το Τμήμα Εσωτερικής ε, Ασφάλειας και θα πρέπει να φροντίσουμε να δοθεί συνέχεια από πλευράς των κρατών μελών που συμμετέχουν και επίσης είναι δική μας ε, ευθύνη ε, να ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας σχετικά με αυτά που μας είπαν οι Αμερικανοί. Άλμπερτ ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ πολύ ε, με τα όσα είπε τώρα μόλι η ρεπόρτα Μετσόλα. σω θα έπρεπε όμω ε, σε, σε μελλοντικέ αποστολέ ε, να φροντίσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για διάφορα σημεία. Αυτό το ε, συνεχέ μέσα έξω από, το, από την κάθε συνάντηση συχνά σημαίνει ότι δεν έχουμε. ότι δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε όσο θέλουμε στις συζητήσεις. Θα ήταν ωραίο να έχουμε περισσότερο χρόνο με τους συνομιλητές μας. Ευχαριστώ και εγώ θα συμφωνήσω. Να ευχαριστήσω όμως ε, και εγώ τη Γραμματεία που οργάνωσε αυτήν την πολύ χρήσιμη αποστολή που κάλυψε ευρύ φάσμα θεμάτων ε, με τα οποία ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή. Εάν ε, δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο για το θέμα αυτό, φτάνω στο τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης, που είναι η ερώτηση επαριθμών επί 005798-16 της κυρίας Ινετφέλτ ε, σύμφωνα με τον κανόνα 134, με το άρθρο 134 του κανονισμού. Ε, ε, σύμφωνα με τον κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει απαντήσει εντός τριών εβδομάδων. Ε, η προθεσμία έληξε στις 31 Οκτωβρίου ε, χωρίς ε, να έχει ληφθεί απάντηση και η κυρία Ινετφέλτ ζήτησε να τεθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνάντησης, ε, της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, σύμφωνα με, τον, με το άρθρο 130, παράγραφος 4 του κανονισμού. Κυρία Ινετφέλτ, νομίζω ότι είναι σημαντικό θέμα και είναι κρίμα που συζητιέται ε, τώρα στο τέλος ε, τη συνεδρίασής μας, βέβαια τελευταία στιγμή μπήκε και στην ημερήσια διάταξη, έχει να κάνει με τις ε, κατηγορίες ότι η Yahoo ε, διάβαζε, εξέταζε τα email των πελατών της για τις κρατικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών όπως είχαν ζητήσει ε, οι υπηρεσίε πληροφοριών ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ σημαντικές κατηγορίες αυτές ε, και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει εάν γνώριζε τις κατηγορίες αυτές, εάν έχει ζητήσει διευκρινήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε τις δραστηριότητες αυτές όταν υιοθετήθηκε το Privacy Shield και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Yahoo έχει παραβεί τους κανόνες περί ασφαλούς λιμένα. Και εάν θεωρεί ότι αυτές οι δραστηριότητες ε, θα είναι ε, ε, νόμιμες υπό το Privacy Shield. Νομίζω ότι είναι πολύ σκόπιμες οι ερωτήσεις αυτές. Εδώ ότι και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν την Yahoo και ότι διαπραγματευόμαστε καλή την πίστη με τις ΗΠΑ όπως είδαμε κατά την προηγούμενη συζήτηση. Με εκπλήση, λοιπόν που δεν απάντησε πάρα πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ακόμα περισσότερο με εκπλήση, ότι ο κύριος Τζανκαρέλη μόλις αποχώρησε. Αναρωτιέμαι τι έχει να πει η Επιτροπή. Διότι συχνά όταν ε, ε, θέτει κανείς τέτοιες ερωτήσεις ε, κατηγορείται ότι είναι αντιαμερικανός. Σε αντίθεση με τα όσα πιστεύει ο κύριο Τραμπ, εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι μεγάλη σημαντική χώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Με ενδιαφέρουν όμω και τα δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρω ότι δεν πρέπει να πυροβολήσουμε τον ε, τον ε, ταχυδρόμο, ε, αλλά περιμένω να ακούσω τι έχετε να μου πείτε. Ε, ναι, η απάντηση βρίσκεται στα τελευταία στάδια της γραπτής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λογικά θα σταλεί την Παρασκευή στο Ευρωκοινοβούλιο η κυρία Νετφέλε. Ευχαριστώ, ενδιαφέρον αυτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μία ερωτήση, ερώτηση στην οποία θα μπορούσε να μας απαντήσει αμέσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αν γνώριζε την κατάσταση αυτή κατά τις διαπραγματεύσεις του Privacy Shield. Αυτό δεν ε, θα πρέπει να απαιτεί ε, συμφωνία από το σώμα των ε, επιτρόπων, αλλά τέλος πάντων θα περιμένουμε την Παρασκευή. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λήξη της συνεδρίασης. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα πραγματοποιηθεί 14 Νοεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και 17 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί.